παρόντες εξ ονόματος της Επιτροπής μας σε συνεργασία σήμερα με τις Επιτροπές Ήτρε, ΑΦΚΟ και Νομικών Υποθέσεων. Συμπροεδρεύει και η κυρία Σπινέλη και η κυρία Φεράρα αντιστοίχω και ο κύριος Κέλλη από την Επιτροπή βιομηχανίας. Επίσης ε, πρώτος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής ΙΜΚΟ, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, και από την Επιτροπή Πολιτισμού η κυρία Φερχάιεν, που εκπροσωπεί τον πρόεδρο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και ελπίζω οι συνάδελφοι να βρουν την διαδικασία ανοιχτή και δημοκρατική Σήμερα έχουμε την πρώτη ακρόαση μια σειρά ακροάσεων μετά από την απόφαση της διάσκεψης των πρόεδρων στις 12 Απριλίου και μετά από μια συνάντηση του κυρίου Ζούκερμπεργκ με την διάσκεψη των πρόεδρων την οποία έχετε δει υποθέτω. Ο σκοπός της σημερινής και των επομένων ακροάσεων είναι κάπως διαφορετικός. Να γίνει δηλαδή μια ακρόαση εις βάθος με τους βασικούς συνομιλητές της και του σκανδάλου. Στόχος είναι να αντλήσουμε διδάγματα και να δούμε το τι θα γίνει στο μέλλον χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάθεσή της. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την υπόθεση και να καταλάβουμε ακριβώ το τι συνέβη, γιατί συνέβη και πώ ε, μπορούσαν να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Η δεύτερη ακρόαση θα γίνει στι 25 Ιουνίου και η τρίτη στις 2 Ιουλίου. Και βεβαίω ε, θα έχουμε και εκπροσώπους του Facebook. Σήμερα δεν έχουμε κάποιον. Συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω βεβαίω τους κανόνε. Απλά πράγματα, μία ερώτηση, αναβουλευτή και μετά μία απάντηση. Πέρα από την συνεδρίαση, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν στην κατανομή των 27 ερωτήσεων και να μας πούν ποιοι βουλευτές θα πάρουν τον λόγο και έτσι έχουμε φτιάξει έναν κατάλογο των ομιλητών. Μετά τις, ε, από τις παρουσιάσεις θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στους Προέδρους των Εν Επιτροπών και μετά θα ακολουθήσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Αλλά και πάλι να σας υπενθυμίσω ότι θα κάνετε μία ερώτηση για ένα λεπτό το πολύ. Θα πείτε σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση δεν κάνετε, μην κάνετε δηλαδή μια γενική ερώτηση, γιατί μία απάντηση θα λάβετε μόνο. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας πείτε σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση και μετά ο κάθε πανελίστας θα έχει δύο λεπτά για να απαντήσει στην ερώτηση. Θα κόβω το μικρόφωνο στο ένα λεπτό. Αν δείτε τον κατάλογο θα μιλήσουμε εξής. Finally, um, I'm going to... είναι στον κατάλογο, δηλαδή Τέλος, θα κάνω την ε, παρουσίαση των ομιλητών. Έχουμε τον κύριο Σάντι Παρακάλης, ε, επικεφαλή Στρατηγική στο Κέντρο για την Ανθρώπινη Τεχνολογία και πρώην διευθυντή επιχειρήσεων του Facebook. Την κυρία Κάρολ Καντουαλντάρ, ε, δημοσιογράφο του Guardian που ερεύνησε την υπόθεση αυτή και την έφερε στη δημοσιότητα, η κυρία Elizabeth Denham, Επίτροπο Πληροφοριών στο ICO του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία συνοδεύει ο κύριος James Dipple Johnston, βόηθος επιτροπός, ο καθηγητής David Carroll, καθηγητής στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ε, ζήτησε από τα Βρετανικά δικαστήρια να αποκαλύψει η Cambridge Analytica πώς συνέταξε το προφίλ του. Και τέλος ο Christopher Wiley, ο οποίος ε, ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε την υπόθεση και πρώην διευθυντής έρευνας στην Cambridge Analytica. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και απαντήσετε τόσο γρήγορα στην, ερώτηση, στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν. Περνάμε τώρα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις των ομιλητών και ξεκινάμε με τον κύριο Σάντι Παρακάλης. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να έρθω να μιλήσω σε εσά σήμερα. Ονομάζομαι σαν αντιπαρακύλες ε, και εργάζομαι για τον μικροδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος εστιάζεται στην επανευθυγράμμιση των ε, συμφερόντων της τεχνολογίας με, αυτόν, με αυτά της ανθρωπότητας. Υπήρξα ε, manager στη Facebook το 2011 και το 2012 και μια από τις κυρίες μου ευθύνες εκείνη την εποχή ήταν η προστασία των δεδομένων σε πλατφόρμες του Facebook. Ήρθα λοιπόν να σας μιλήσω για το τι συνέβη από πλευράς Facebook με την Cambridge Analytica να σας πω τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πριν μπούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς το Facebook ενεπλάκει στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, ήθελα πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα του ε, Facebook. Αυτό πρέπει να καταλάβετε γιατί η πλατφόρμα του Facebook είναι ότι είναι μια υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία και που επιτρέπει σε εξωτερικούς προγραμματιστές, σε εξωτερικές εφαρμογές να δημιουργούν εφαρμογές που αποκτούν πρόσβαση ε, σε δεδομένα του Facebook ε, για χρήστες του Facebook και λειτουργεί και σε desktop ε, και σε υπολογιστή και σε κινητές συσκευές όπως βλέπετε στα δεξιά. Και σε, από υπολογιστέ κανονικού, όπω βλέπετε στα αριστερά, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ένα βασικό κομμάτι της έρευνας βασίζεται στο πώς οι εφαρμογές λαμβάνουν τα δεδομένα από το Facebook. Αυτό είναι βασικό ε, θέμα εδώ πέρα. Κάθε φορά λοιπόν που ένας χρήστης του Facebook θέλει να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή στο Facebook, συμφωνεί σε μια οθόνη συμφωνίας που μοιάζει με αυτήν εδώ, που είναι, χρονολογείται πριν από μερικά χρόνια, αλλά υπάρχουν νεότερες εκδοχές τώρα και μόλις πατήσει allow, επιτρέπεται ο χρήστης, ή συμφωνώ, η εφαρμογή σε αυτή την περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση στο Amazon, λαμβάνει τα δεδομένα του χρήστη όπω προσδιορίζεται στην οθόνη ε, στην οποία πάτησε συμφωνώ ο χρήστη. Πώ λειτουργεί η ροή των δεδομένων πρώτα απ' όλα δίνει τα δεδομένα του χρήστη στο facebook, το όνομά του, άλλε πληροφορίε για τον εαυτό του, ε, μετά ε, συνενεί στο να τα χρησιμοποιεί αυτή η εφαρμογή, στον έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που ονομάζονται και μετά το Facebook διαβιβάζει στην εφαρμογή τα δεδομένα αυτά. Και εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα με την Cambridge Analytica, ότι μόλις η εφαρμογή αποκτήσει στα χέρια της αυτά τα δεδομένα, ουσιαστικά το Facebook δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα κάνει με τα δεδομένα αυτά ο προγραμματιστής της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι αν ο προγραμματιστής είναι κακόβουλος, μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Στη προκειμένη περίπτωση ε, μιλάμε για τον Κόγκαν ως προγραμματιστή και το τρίτο μέρος ήταν η Cambridge Analytica. Το τέταρτο μέρος μάλλον, συγγνώμη. Ε, ένα άλλο πράγμα βασικό πρέπει να καταλάβουμε είναι πώς οι προγραμματιστές μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς ρητή συνένεση των χρηστών. Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ε, μέχρι το 2014, ουσιαστικά μέχρι το 2015 σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εφαρμογές του Facebook μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε δεδομένα των χρηστών των ανλόγων εφαρμογών, αλλά και δεδομένα των φίλων των χρηστών. Κατά μέσο όρο, ε, ένας χρήστης του Facebook έχει 200 με 300 φίλους. Υπάρχει τεράστια ε, μεγέθυνση λοιπόν των δεδομένων που λαμβάνει μια εφαρμογή όταν χρησιμοποιήσει τους φίλους ενός ε, χρήστη της. Και έχουμε μια νέα ιστορία που σήμερα δημοσιεύτηκε, σήμερα το πρωί στην New York Times. Μπορείτε να μου κάνετε ερώτηση για αυτήν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Ε, και για το αφορά του κατά πόσο συνεχίζεται αυτό ή όχι. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα ίδια τα δεδομένα. Πολλά λοιπόν δεδομένα μπορούν να λάβουν οι προγραμματιστές από το Facebook. Εδώ βλέπετε μια λίστα ορισμένων πραγμάτων που υπήρχαν πριν από την αλλαγή του 2014. Μπορείτε να δείτε δηλαδή ότι οι προγραμματιστές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πράγματα όπως τις δράσεις ενός χρήστη, ε, αναρτήσεις του χρήστη, πιο ευαίσθητες πληροφορίες, ε, σχέσεις, ε, θρησκεία, πολιτικές πεπιθήσεις. Όλα αυτά μπορούσαν να τα δουν και για τους φίλους τους. Και υπήρχαν και εκτεταμένα δικαιώματα που έδιναν στους προγραμματιστές ακόμη περισσότερη πρόσβαση σε δεδομένα για παράδειγμα, η επέκταση αυτή των δικαιωμάτων μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να διαβάσει και ιδιωτικά μηνύματα. Τι ε, έγινε λάθος λοιπόν με την Cambridge Analytica και το Facebook. Πρώτα απ' όλα το Facebook δεν είχε καμία δυνατότητα να παρακολουθεί ούτε να ελέγχει τη χρήση των δεδομένων αφού τα είχε διαβιβάσει στους προγραμματιστές εφαρμογών. Δεύτερον, έδωσε τη δυνατότητα σε εφαρμογές να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα φύλων χωρίς ρητή συνένεση. Τρίτον, ε, ε, έκαναν ελάχιστο έλεγχο ή καθόλου έλεγχο για τους προγραμματιστές. Τέταρτον, ε, στην περίπτωση της Cambridge Analytica βασίστηκαν στην υπόσχεση του προγραμματιστή ότι διαγράψει τα δεδομένα. Και έκαναν μηνύσεις αφού μόνο αποκαλύφθηκε η κατάχρηση. Και τέλος, το Facebook δεν απογράψει στην Cambridge Analytica να αναρτά διαφημίσει στο Facebook μετά από την πρώτη του ε, δράση το 2000, στα τέλη του 2015. Η Cambridge Analytica λοιπόν συνέχισε να ε, κάνει διαφημίσει στο Facebook για άλλα δύο χρόνια, μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Οπότε ε, πολλά στοιχεία χαρακτηρίζουν αυτό το συγκεκριμένο θέμα αλλά ένα που ήθελα να τονίσω είναι ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ ευρύτερο από το Facebook και την Cambridge Analytica. Εδώ σε αυτό το την απέσια εικόνα, την τρομακτική εικόνα. Βλέπετε τη διαφημιστική βιομηχανία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ βλέπετε σε κάθε λογότυπο κάποια εταιρεία που με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην μετατροπή των δεδομένων χρηστών σε χρήματα. Φανταστείτε να προσπαθείτε να ρυθμίσετε όλη αυτή την πολύπλοκη βιομηχανία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Η καλή είδηση είναι ότι το GDPR είναι ένα πρώτο καλό βήμα για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των χρηστών. Αλλά όπως ανέφερα, είναι εξαιρετικά περίπλοκο το πρόβλημα. Ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω τέσσερα πράγματα που θα σας επισημάνουν τι πρέπει να δείτε ουσιαστικά σε περίπτωση που αποφασίσετε περαιτέρω ρυθμίσει, περαιτέρω νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει κατανόηση και όχι απλά συνένεση. Εδώ στην εικόνα αυτή. Βλέπετε τους όρους χρήσης, ε, ε, την οθόνη ε, συμφωνίας που χρησιμοποιεί το Facebook και που λέει ότι συμφωνεί με το GDPR. Σας επισημαίνω ότι τα links εδώ που υπάρχουν για να διαβάσει κανείς τους όρους χρήσης και για να δει τις επιλογές που έχει είναι με πάρα πολύ μικρά χράματα και το κουμπί δέχομαι accept για να χρησιμοποιήσει κανείς το Facebook αμέσως είναι τεράστιο σε σχέση με την υπόλοιπη σελίδα. Οπότε η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο χρήστη να ενθαρρυνθεί να δεχθεί τα πράγματα χωρί περαιτέρω δράση. Θέλουμε εμεί να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστε αντιλαμβάνονται σε τι συμφωνούν. Ότι δεν απλά συνενούν, δεν δέχονται απλά χωρί να έχουν διαβάσει ε, τι, τι ακριβώ, σε τι ακριβώ έχουν συμφωνήσει. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπου να ευθυγραμμίσουμε ε, κίνητρα για τι επιχειρήσει και για του χρήστε. Και μια πολύ καλή ε, μεταφορά εδώ είναι η παρομοίωση είναι η σύγκριση συγγνώμη, είναι οι ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε η υλοποίηση των ε, ζωνών ασφαλείας δεν βασίστηκε σε αποφάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά σε κίνητρα που είχε η... ο τομέας των ασφαλίσεων. Οι, ασφαλι... οι ασφαλιστικές εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν τεράστιες αποζημιώσεις σε κάθε περίπτωση τραυματισμού. Οπότε αυτού συνέφερε οικονομικά η ασφάλεια των επιβατών των αυτοκινήτων. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε με την προστασία των δεδομένων. Ουσιαστικά, αν φτιάξουμε ένα στιβαρό ε, πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ε, μπορούμε να οθήσουμε ε, το τομέα της ασφάλειας με τον παρόμοιο τρόπο ώστε να εκπαιδεύσει χρήστες και εταιρείε για τις βέλτιστες πρακτικές και έτσι να κατανεμηθεί ο κίνδυνο ε, σε πολλέ εταιρείε όσον αφορά τι κυρώσει και τι ποινέ, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε φορά που υπάρχει μια πετρελαϊκή κοιλίδα, για να την πούμε έτσι, δεν θα πληρώνεται από μια εταιρεία μόνο, αλλά θα κατανέμεται το κόστο ε, σε, σε, σε, σε πολλού τομεί. Το τρίτο που ήθελα να αναφέρω αφορά την προγραμματική πρόσβαση σε δεδομένα για του χρήστε. Όπω και με την ασφάλεια, πρέπει να δημιουργήσουμε εταιρείε που να τη συμφέρει να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των χρηστών και την προστασία των δεδομένων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε. Οι κανόνε από μόνοι του δεν λειτουργούν. Θέλω να σα δείξω λοιπόν ένα προσωπικό παράδειγμα. Εδώ βλέπετε το ιστορικό των ερευνών των δικών μου στο Google πριν από 8 χρόνια. Ε, τα έχει ακόμα η Google. Το παρατήρησα γιατί πήγα στο εργαλείο My Activity, η δραστηριότητά μου, και μου έκανε έκπληξη και ενοχλήθηκα κάπω που ακόμα έχουν αυτά τα στοιχεία αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι θα μπουν στον κόπο να πάνε να διαχειριστούν όλα τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι εταιρείε για αυτού, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το κάνει κανεί σε όλε τι υπηρεσίε που χρησιμοποιεί. Αν λοιπόν εφαρμόσουμε την απέτηση να υπάρχει προγραμματική πρόσβαση για όλα αυτά τα δεδομένα και τι λειτουργίε, θα δημιουργήσουμε νέε εταιρείε οι οποίε θα βοηθήσουν του χρήστε στη διαχείριση δεδομένων του. Είτε μιλάμε για τα βασικά του δεδομένα, ή για να τους βοηθήσουν να συγκεντρώσουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν αλλού ε, εφόσον το επιλέξουν. Το τέταρτο που ήθελα να επισημάνω, τέλος, είναι ότι καθώς ε, προετοιμαζόμαστε για να εκπονήσουμε νέους κανονισμούς, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου την προστασία των μικρών εταιριών, οι οποίες ε, είναι η κινητήρια δύναμη της καινοτομία ε, σε όλους τους τομείς. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πολύ καλά το πώς θα τις βοηθήσουμε να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες και πώς αυτοί οι νέοι κανόνες θα τις επηρεάσουν. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ε, ενδυναμώσουμε περαιτέρω τα μονοπόλια μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων. Και τέλος ήθελα να πω ο κόσμος είναι στραμμένος προς εσάς. Σε εσάς απευθύνεται για την νομοθεσία, για τους κανονισμούς, για την προστασία δεδομένων. Και να είστε βέβαιοι, πολλοί Αμερικανοί θέλουν να υπάρχει κάτι στι ΗΠΑ όπω το GDPR και οι περισσότεροι υπάλληλοι ε, τεχνολογικών εταιριών που γνωρίζω εγώ ε, το ίδιο ελπίζουν και θα σας θαυμάζουν για το GDPR. Σας συγχαίρω λοιπόν και ελπίζω να συνεχίσετε τη δράση σας ε, και την καινοτομία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μητέρα της GDPR είναι εδώ, ο πατέρα, δεν ξέρουμε που είναι. Ε, δεν σας πληρώσαμε εμεί για τα καλά σας λόγια, το διευκρινίζω αυτό. Και να πω ότι όλοι εδώ πέρα ε, από όλου τους μιλητέ μας ζητήσαμε μια παρουσίαση μέχρι 10 λεπτά. Λοιπόν, ακολουθούμε τώρα την Κάρολ Καλτγούλντερ, δημοσιογράφο στην Guardian που ερεύνησε την υπόθεση αυτή και συνεχίζει να ασχολείται με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε και χαίρομαι ιδιαίτερος που κάνετε αυτές τις ακροάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές θεωρώ και επίγουσες ε, και πραγματικά απαιτείται ε, σοβαρότερη εξέταση των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να απαντήσουμε ως δημοσιογράφοι. Εγώ ερευνώ αυτά τα ζητήματα τώρα εδώ και 18 μήνες και μπορούσα να, θα μπορούσα να σας πω διάφορα, αλλά θα ήθελα να εστιάσω στο εξής. Ε, το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορες έρευνες αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την εκστρατεία για να φύγουμε από την Ένωση. Ο Επίτροπος Πληροφοριών Έρευνα, η Εκλογική Επιτροπή επίσης. Υπάρχει μία έρευνα από την αστυνομία ε, από το Κοινοβούλιο υπό την προεδρία του Ντέμιαν Κόλλινς που εξετάζουν πιθανά αδικήματα όπως ε, υπερβολικές ε, δαπάνες, παράνομος διαμοιρασμός δεδομένων, πιθανή διαγραφή στοιχείων, παράνομος συντονισμός των εκστρατιών. Να σας ενημερώσω λοιπόν πώς έχουν οι νόμοι μας περί εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ελέγχουμε τις δαπάνες τις διαφημιστικές και αυτό θα έλεγα είναι το θεμέλιο τη δημοκρατική διαδικασία. και η νομοθεσία αυτή έχει αναπτυχθεί σταδιακά επί 100 χρόνια και αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι ψηφιακές εκστρατείες έχουν αλλάξει τη λειτουργία της νομοθεσίας. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον οι νόμοι αυτοί δεν λειτουργούν και αυτό θεωρούν διάφοροι νομικοί και πανεπιστημιακοί. Τώρα περνάνε όλα μέσω των τεχνολογικών εταιριών και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Οπότε αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν στο δημοψήφισμα, ποιος τα ξόδεψε, από πού ήρθαν, ε, τι διαφημίσεις είδε ο κόσμος, πώς ε, έγινε η στόχευση, τι, ε, σε τι δεδομένα βασίστηκαν. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στους ε, σερβερ του Facebook και της Google, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόσβαση. Οπότε έχουμε την εξή κατάσταση. Έχουμε ξένες εταιρείε που έπαιξαν κέριο ρόλο σε μια κέρια εκλογική διαδικασία και δεν έχουμε κάποιον τρόπο για να αποκτήσουμε αυτές τις πληροφορίες να σα πω πω αισθάνεται ένα δημοσιογράφο που προσπαθεί να βρει απαντήσει Είναι σχεδόν αδύνατον. Ο Guardian ανέφερε πρώτη φορά τα τη Cambridge Analytica και τη συλλογή δεδομένων τον Δεκέμβριο του 2015. Ο Χάρι Ντέιβι ασχολήθηκε με το θέμα. Και τα ξέραμε και τότε αρκετά από αυτά τα πράγματα. Ο Χάρη πήγε στο facebook και έκανε πολλέ ερωτήσει, αλλά απαντήσει δεν έλαβε. Κατόπιν ήρθαν. Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν και αυτοί το ρεπορτάζ ο κύριος ε, Στρέσαντζερ στην Ελβετία, ο Χάρι Σουόρτς επίσης ε, και εγώ. Και κάνουν ό,τι θέλουν αυτές οι πλατφόρμες, αποφεύγουν τις απαντήσεις. Στην περίπτωσή μας μας απείλησαν κιόλας ε, κατά κάποιον τρόπο και όταν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα έχουμε κάποια μερική πληροφόρηση. Ο Σάντι ανέφερε ότι εμφανίστηκε χτες μια ιστορία στους New York Times όπου μάθαμε ότι οι απαντήσεις ε, του Μάρκ Ζουκερμπέκ στο Κογκρέσο δεν ήταν παραπλανητικές αλλά ήταν τουλάχιστον ελλειπείς. Οπότε εσείς είστε θα έλεγα το θεσμικό όργανο που έχει το ανάστημα να σταθεί απέναντι σε αυτούς τους τεχνολογικούς γίγαντες και μόνο εσάς φοβούνται θα έλεγα. Ε, ελπίζω πραγματικά να τους κάνετε να λογοδοτήσουν κάτι το οποίο δεν είδαμε όταν ήρθε εδώ ο Μάρκ Σούκερμπεργκ. Έχω την εντύπωση ότι του επετράπει να εμφανιστεί συνεργάσιμος χωρίς να είναι συνεργάσιμος. Κλασικό δηλαδή για τον Ζούκεμπεκ. Να σας πω λοιπόν πώς μπλέκτηκα εγώ σε αυτήν την ιστορία. Το Δεκέμβριο του 2016 άκουσα για πρώτη φορά για την Cambridge Analytica από έναν Αμερικανό πανεπιστημιακό όνομα τη Jonathan Albright. Έγραψα ένα άρθρο και... Ε, έλεγα ότι δούλευαν για την εκστρατεία του Τραμπ και για την εκστρατεία του να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λένε δεν εργαστήκαν ποτέ σε κάτι τέτοιο. Αλλά υπήρχαν τα στοιχεία στο site live.eu λένε είχαμε προσλάβει την Cambridge Analytica. Οπότε απευθυνθήκα σε έναν επιχειρηματία ο οποίος ήταν από τους κύριους χρηματοδότες και του Νάιτζελ Φάρατζ και της εκστρατείας και ο Νάιτζελ Φάρατζ είναι βεβαίως βασική μορφή τη υπόθεση και ελπίζω να του κάνετε ερωτήσει ε, που δεν ε, έχουν γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Φάρα Τζέφερε σε επαφή την Cambridge Analytica με την έξτρατη ε, αυτή λόγω της φιλίας του με τον Ρόμπερτ Μέσερ και τον Στίβ Μπάνον. Οι δύο αυτοί με τη σειρά τους έπαιξαν κέριο ρόλο στην υπόθεση αυτή πέρα από την στήριξή τους στην εκστρατεία έφεραν και το site Breitbart στο Ηνωμένο Βασίλειο που στήριξε επίσης την εκστρατεία του Νάιτζελ Φάρατ για να φύγει η Μεγάλη Βρετανία και ο Ντάντι Βουίκα μου είπε ότι και αυτό το έχω ηχογραφημένο πριν να αρχίσουν οι διαψεύσεις ότι η Cambridge Analytica τους βοήθησε δωρεάν. Δεν τους κλήρωσαν γιατί είχαν λέει τους ίδιου στόχους όπως είχαν και στις ΗΠΑ. Ε, Υπήρχε μια φιλία μεταξύ των Μπάνων, Μέρσερ και Φάραντς και είπε ότι τους βοήθησαν να καταλάβουν τι έκαναν με τα δεδομένα του Facebook, πώς να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές δεδομένων, πώς να χρησιμοποιήσουν τα συναισθήματα, τον φόβο για να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί αναλόγως. Ε, σύντομα λοιπόν ε, θα περάσω στα επόμενα βήματα. Μετά από αυτή την ε, δωρεά, η δωρεά αυτή είναι πιθανώς παράνομη και έπρεπε να δηλωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξεκίνησαν δύο έρευνες, ε, τη μία θα σφεί η κυρία Αντέναμ, αλλά αμέσως μετά μου έγραψε ένας αναγνώστης από τον Καναδά και μου είπε ότι η Cambridge Analytica είχε υποκατάστημα στον Καναδά, SAR Canada λεγόταν, και πεσήμανε ότι ο διευθυντής του υποκαταστήματος ήταν επίσης διευθυντής μιας άλλη εταιρεία ονόματι Aggregate IQ η οποία συνεργαζόταν με μια άλλη εκστρατεία, την επίσημη ας πούμε εκστρατεία, το Vote Leave και με τρεις άλλες ε, εκστρατείε, με το DUP, με τους Βετεράνου για την Βρετανία και με το ΛΥΠ. Και έχουμε πολύ αυστηρού ε, νόμους όσον αφορά τον συντονισμό διαφόρων προεκλογικών εκστρατιών. Κάτι το περίεργο λοιπόν συνέβαινε εδώ, είχαμε μια υπόγεια σύνδεση και μόλις ρώτησα κάτι για την Cambridge Analytica έσβησαν τις σχετικές λεπτομέρειες από την σελίδα τους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι ε, το οποίο γινόταν ε, εγκρυπτό. Και βεβαίω εδώ πέρα μίλησαν και οι πρώην υπάλληλοι, τους οποίους ευχαριστώ και ο κύριος Βάλλη, ο οποίος ε, θα σας πει σε λίγο τα πράγματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Για να συνοψίσω λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ο Μάρκ Ζούκερμπερ και σας είπε, κάναμε λάθη, αντλήσαμε τα διδάγματά μας, περισσότερη διαφάνεια στο μέλλον. Αυτό λέει πάντα το Facebook, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να μάθουμε τι έγινε στο παρελθόν. Πρέπει να μάθουμε το τι συνέβη στο δημοψήφισμα και τι λεφτά ξοδεύτηκαν από ποιον και εάν αυτό έγινε νομίμως και ότι ε, έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να διακριβωθούν τα ακριβή γεγονότα. Υπάρχει ένας κίνδυνος λοιπόν μιας συστημικής αποτυχίας σχεδόν, αυτό το οποίο είδαμε δηλαδή στην Βρετανία, στο δημοψήφισμα, γιατί είμαστε σε μια θέση όπου ε, δεν λειτουργήσε η εκλογική νομοθεσία, δεν μπόρεσε να το προλάβει αυτό το φάσμα αυτό ενεργειών και γνωρίζουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές ε, και ειδικά η Εκλογική Επιτροπή δεν είχε το νομοθετικό πλαίσιο ε, που χρειαζόταν και δεν είχε και τις αρμοδιότητες για να ζητήσει τα στοιχεία. Επίσης ξέρουμε ότι είναι πια αργά το ε, site ε, live.eu πλέον έχει παραπεμφθεί στην αστυνομία, αλλά είναι δύο χρόνια μετά το γεγονό ε, και βέβαια οποιαδήποτε δίκη θα είναι κατόπιν εορτή, αφού έχει φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει και μια πολιτική αποτυχία εδώ και αστοχία, γιατί δεν είναι μόνο η η κυβέρνηση η οποία θέλει το Brexit με κάθε κόστος και πραγματικά δεν βλέπει. Αλλά πιθανώς ε, έχει και κάποια συνενοχή, γιατί δύο υπουργοί της νυν κυβέρνησης, ο Μάικλ Γκόβ και ο Μπόρις Τζόνσον, ήταν διευθυντές ε, της εκστρατείας Vote Leave και ε, είναι πιθανόν να είχαν πλήρη γνώση των υπερβολικών δαπανών. Ε, δύο πολιτικοί διευθυντές της Τερέζας Μέη έχουν κατονομαστεί ως άμεσα υπεύθυνοι για τις υπερβολικές δαπάνες. Οπότε Πραγματικά προβληματίζομαι και με συγχύζει το γεγονός το ότι ίσως δεν έχουμε κράτος δικαίου στην Βρετανία όσον αφορά την εξαγωγή του δημοψηφίσματος και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε τα πράγματα από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Um... Ευχαριστώ πολύ. Κάρολα. Επίσης, ε, στην καρδιά τη έρευνα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με την Cambridge Analytica ήταν ε, ο, η Επίτροπος Elizabeth Dennon, μόλις την ανέφερε η Κάρολ. Αλλά είμαι ευτυχής που δέχτηκε την πρόσκληση, γιατί έτσι θα έχουμε πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ελίζαμπεθ Ντένον, παρακαλώ λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, αξιότιμη κυρία Προβλεφτές, που με καλέσατε στη σημερινή ακρόαση. Εγώ είμαι επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου για την ε, ε, ενημέρωση και δεσμεύομαι από την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το γραφείο μου, που είναι γνωστός ICO, είναι νομίζω η μεγαλύτερη αρχή προστασίας δεδομένων στην Ένωση όσον αφορά αριθμό προσωπικού και ε, χρηματοδότηση. Είμαστε ένας ενεργός ε, νομοθέτη, ε, ρυθμιστής, μάλλον έχουμε ρόλο πέρα από την ανάθεση, μάλλον την διερεύνηση καταγγελιών σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα για το θέμα αυτής της ακρόασης η υπηρεσία μου ηγείται της έρευνας για το Facebook και την Cambridge Analytica εξ ονόματος των εταίρων μας της Ένωσης των ομολόγων μας της Ένωσης. Κάποιες άλλες επίσης ε, εθνικές αρχές έχουν ε, διενεργήσει έρευνες σε σχέση με διάφορες νόμιμες ανησυχίες σε σχέση και καταγγελίες σε σχέση με το Facebook. Με συνοδεύομαι δε από τον ε, αναπληρωτή επίτροπο James Dipple Johnson, ο οποίος ηγείται των επιχειρήσεων στο γραφείο, του, του, γραφείου μου, καθώς και διενεργεί και έχει μάλλον λάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνά μας για τη χρήση των αναλυτικών δεδομένων για πολιτικούς τους σκοπούς ή οι πολιτικές εκστρατείες. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα η τυπική έρευνα η επίσημη έρευνα και γι' αυτό και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορούμε να πούμε και ίσως σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μου υποβάλλετε να μην μπορώ να απαντήσω. Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση σε σχόλια που έκαναν άλλοι ομιλητές. Με τα χαράς θα απαντήσω λεπτομερώς στην Επιτροπή σας γραπτός όταν θα είμαι σε θέση να αποκαλύψω άλλες πληροφορίες, περαιτέρω πληροφορίες. Καταρχάς θα ήθελα όμως να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και το κοινό που ίσως παρακολουθεί ότι κατανοώ την ε, ε, δύσκολη θέση ή την ανησυχία σε σχέση με το, την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα και με ποιον τα μοιράζεται αυτά. Πρόσφατα είδαμε ότι το σύστημα αυτό έχει εφαρμοστεί στις πολιτικές εκστρατείες για να επηρεάσει το πώς ψηφίζουμε και ανησυχώ ιδιαίτερα για το ότι αυτό συνέβη χωρίς την κατάλληλη νομική ή ηθική ε, κάλυψη για τον αντίκτυπο που έχει αυτό στο δημοκρατικό μας σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει πως το επιγραμμικός χώρος είναι τελείως ε, αρρύθμιστος ή απορριθμισμένος. Οποτεδήποτε επιγραμμικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, τότε η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται και μπορεί να παρέχει αποτελεσματική προστασία για, τους, ε, για τα άτομα. Η προστασία δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα στον Ευρωπαϊκό Χάρτη και το, το ΔΕΚ και η νομολογία το έχουν καταστήσει σαφές ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ελέγχουν τα δεδομένα ε, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασία δεδομένων. Μπορεί δηλαδή να, είναι, ε, να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ε, κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν έλεγχο για το τι συμβαίνει, ελέγχουν το τι συμβαίνει για τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ανθρώπου, μπορούν να διλύσουν το περιεχόμενο, ελέγχουν τι βλέπουμε για να μπορούμε να το δούμε και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ε, είναι αυτοί που τους αποφασίζουν. Οι online πλατφόρμες δεν μπορούν να λένε πως είναι απλά πλατφόρμες για το περιεχόμενο. Πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προέλευση της πληροφορίας που ε, παρέχουν στους χρήστες. Ωστόσο αναγνωρίζω ότι κάποιες στοιχεία των νομικών μας συστημάτων δεν έχουν μπορέσει να συμβαδίσουν με την απρόβλεπτο ρυθμό της ανάπτυξης του ίντερνετ. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων και τη σχετική νομοθεσία, το GDPR είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ε, νομοθεσία, αλλά και μεγάλο βήμα όσον αφορά τις αρχές προστασίας δεδομένων. Το GDPR έχει γραφτεί ευέλικτα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι υποπτικές αρχές όπως η δική μου ICO θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα δεδομένα και να βλέπουν ε, και να αποφασίζουν ποιος είναι ο ελεγκτής των δεδομένων άσχετα από το μέσο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων και η πρόσβαση σε μια αρχή εποπτική για τα δεδομένα ε, πηγαίνει πολύ πιο πέρα από ένα απλό γραφείο. Τα, τα, τα εγκλήματα, τα αδικήματα μάλλον που αφορούν δεδομένα είναι πραγματικά αδικήματα και αυτό ε, ακόμα και αν ε, η παρανομία έχει συμβεί πλήρως online. Όπως ίσως πολύ γνωρίζετε, το Μάιο του 2017 ανακοίνωσα επίσημη έρευνα εξηγώντας τις ανησυχίες μας σε σχέση με αόρατη επεξεργασία τους αλγοριθμούς, της αναλύσης, ε, την αντιστοίχηση δεδομένων και τα ε, προφίλ που ε, περιέχουν προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούν πολιτικά δεδομένα σε πολιτικές εκστρατείες και εκστρατείες δημοψηφισμάτων. Το Φεβρουάριο του 2018 εστιάσαμε την προσοχή μας στο Facebook και την Cambridge Analytica. Μόνο μία πτυχή της συνολικής μας έρευνας, αυτή λοιπόν εντάθηκαν από τις ε, μαρτυρίες που μας έδωσε ο κύριος Βάιλι, τον οποίο θα ακούσετε σε λίγο. Και ε, με αυτό το υπόβαθρο πολύ έντονου ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτικού κόσμου, ε, εμείς ε, συνεχίσαμε την έρευνά μας. Επίσης δώσαμε ε, μαρτυρία στην, ε, στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διερευνεί σε ψευδείς ειδήσει, fake news, τις οποίες προεδρεύει ο Ντάμιον Κόλλινς ακολουθήσαμε μια διπλή προσέγγιση. Η πρώτη είναι να διερευνήσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες και να καταλήξουμε σε ενέργειες επιβολής του νόμου. Επίσης, δεύτερος άξονας ήταν να εκπονήσουμε έκθεση για τις ευρύτερες επιπτώσεις αυτής της έρευνάς μας, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων όσον αφορά τα κενά της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και αλλού. Και σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε αυτή μας την έκθεση στα τέλη του μήνα. Η έρευνά μας είναι πολύ μεγάλη μεγάλη και ευρύτατη. Έχουμε 40 ερευνητέ που εργάζονται full time η αυτή μα την έρευνα. Ε, συν μια ειδική ε, μονάδα εντοπισμού στοιχείων και ανάκτηση στοιχείων, δηλαδή ακόμα 20 ανθρώπους. Εξετάζουμε πάνω από 20 ξεχωριστούς οργανισμούς, ε, κοινωνικές ε, πλατφόρμες, μεσίτες δεδομένων, εταιρείες ανάλυσης, πολιτικά κόμματα, ομάδες πολιτικών εκστατιών και πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ιδρύματα. Ε, φυσικά πρέπει να ανταποκριθούμε στα πολιτικά και ποινικά στάνταρ συλλογής των μαρτυριών και των ε, αποδεικτικών στοιχείων εάν ε, θέλουμε να χρησιμεύσουν σε κάτι. Έχουμε εκατοντάδες τεραμπάιτ δεδομένων που πρέπει πολύ προσεκτικά να αναλυθούν και αυτά προέρχονται από έρευνες σε διάφορους ε, χώρους και διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά. Έχουμε χρησιμοποιήσει τις ε, αρμοδιότητές μας ε, τα, που περιλαμβάνουν και την ε, ενέργεια κατόπιν εντάλματος. Βλέπουμε μια ολόκληρη σειρά επίσης κυρώσεων που έχουμε στη διάθεσή μας ε, και μπορούμε να υποχρεώσουμε στην παράδοση των αποδεικτικών στοιχείων αλλά και να σφραγίσουμε ψηφιακές ε, μαρτυρίες ή στοιχεία όταν δεν μπορούμε να τα ανακτήσουμε άμεσα. Η έμφαση λοιπόν προφανώς είναι στην προστασία των δεδομένων και να γνωρίζω την μεγάλη σημασία της εργασίας που υπό εξέλιξη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να διασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε στους πολίτες της Ένωσης ότι ε, αν τα, τα δεδομένα τους έχουν ε, ε, πέσει θύματα κακοδιαχείρισης υπάρχει νομική και ρυθμιστική απάντηση που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους προστατεύσει. Τα θέματα που ανέκυψαν μέσω της υπόθεσης Facebook Games Analytica ξεπερνούν την εντολή του ICO εμείς προβαίνουμε σε συστάσεις στην επερχόμενη μας έκθεση που, συστάσεις που ξεπερνούν τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα από την προστασία των δεδομένων, αναμένω η έκθεσή μου να χρησιμοποιηθεί και από άλλους ρυθμιστές που εποπτεύουν εκλογικέ διαδικασίες, αλλά και όσοι ασχολούνται με την ακαδημαϊκή έρευνα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και να ενταθεί η συνεργασία στους τομείς αυτούς. Το κύριο μου μήνυμα για τους ευρωβουλευτές είναι να δώσουν στο GDPR κάποιο χρόνο για να να λειτουργήσει. Η έρευνα του ICO είναι σε τέτοια κλίμακα που είναι άνευ προηγουμένου. Πιστεύουμε πως είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει ποτέ ξεκινήσει από μια αρχή προστασίας δεδομένων. Η έρευνά μας ε, ε, δίνει μια ευκαιρία να εξεταστεί το GDPR και να δούμε αν θα σταθεί απέναντι στις πιέσεις και τις απαιτήσεις μιας πραγματικής σύγχρονης υπόθεσης. Η έρευνά μας και η δράση μας σε αυτή την υπόθεση θα αλλάξει σίγουρα την ε, συμπεριφορά και τη συμμόρφωση όλων των φορέων στο χώρο των πολιτικών εξατειών. Οι δημοσιογράφοι, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, οι υποστηριχτές, οι ε, οι νομικοί σύμβουλοι και οι βουλευτέ έχουν παίξει ρόλο κλειδί στο να φέρουν αυτό το θέμα στην προσοχή του κοινού. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια, ε, μια σταθερή βούληση των πολιτών να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε αρχές προστασίας δεδομένων που δεν θα φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που στη διαθεσή τους και να επιβάλλουν κυρώσεις και πρόστιμα και νομοθέτες που θα στηρίζουν τις αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί πω θα έχουν τη δυνατότητα και την ε, πρακτική ε, εφαρμογή των, του ρόλου τους ε, είμαι ευτυχή λοιπόν που συμμετέχω και απαντώ ερωτήσει, αλλά θέλω να ζητήσω την Επιτροπή σα να σκεφτεί ότι είμαστε στην υποεξέλιξη σημαντική ποινική έρευνα που ξεπερνά την Cambridge Analytica και το Facebook και αυτό μπορεί να περιορίσει κάποιους, τη δυνατότητά μου να απαντήσω και να σχολιάσω κάποια πράγματα. Ευχαρίστω θα ενημερώσουμε τι επιτροπέ του Ευρωκοινοβουλίου σε περαιτέρω φάση εάν ε, υπάρξουν τέτοιε εξελίξει που να μα το επιτρέψουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαστε ιδιαίτερα για όσα είπατε και για τους περιορισμούς. Κύριε καθηγητά, κύριε David Κάρολ, εσείς στραφήκατε στα Βρετανικά δικαστήρια ώστε να υποχρεωθεί η Cambridge Analytica να σας στείλει το ε, προφίλ που είχαν ε, διαμορφώσει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ πέρα ε, να συμμετέχετε στην συνάντηση αυτή. Έχετε το λόγο κύριε Κάρολ. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων για την πρόσκληση της άλλης Επιτροπής και ευχαριστώ ιδιαίτερο τον Δ. Πολ Ολίβιερ Ντεχέι που με συνέστησε αλλά και με βοήθησε να ξεκινήσω την αναζήτηση αυτή για τα δεδομένα μου που με έφερε εδώ σήμερα. Μου δίδαξε πώς ε, τα δεδομένα, η τεχνολογία και η νομοθεσία προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία βοηθούν στην προστασία των δημοκρατιών του 21ου αιώνα. Ε, για να δω αν τα δεδομένα μου ως ψηφοφόρου ε, θα μπορούσαν, είχαν πάει κάπου Εγώ συμβουλεύτηκα τους ε, δικηγόρους μου για το θέμα της Cambridge Analytica για να δω τι έχουν αυτά τα δεδομένα ε, θεωρώντας ότι ήταν αδύνατο να υπάρχει πλήρες αρχείο των δεδομένων μου ως ψηφοφόρου και εγώ ως Αμερικανός πολίτης είχα δικαίωμα Υπέβαλα λοιπόν μια επίσημη καταγγελία ε, στις 4 Ιουλίου του 2017 που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας μάλιστα περιπτώντας στις Πολιτείες. Ε, εκεί αναφέρω ότι ανεπαρκώς ε, έμαθα πώς το προφίλ μου χρησιμοποιήθηκε και τι πληροφορίες δόθηκαν σε τρίτους. Και μετά από την καταγγελία μου, ε, ε, με την καταγγελία μου βοηθήθηκε η έρευνα ε, επί των πρακτικών ανάλυσης ψηφοφόρων. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ με την Επίτροπο Πληροφοριών. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που τη συναντώ αυτό προσώπος. Χαίρομαι για την υποστήριξη και την αναγνώριση της γενικής έννοιας της κυριαρχίας των δεδομένων διότι τα δικά μου δεδομένα υπέστησαν επεξεργασία στον Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ απέδειξα μέσω του Subject Access Request ότι η νομοθεσία πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως υπηκότητας. Η εντολή ε, ε, της ICO ε, έπρεπε να εφαρμοστεί σήμερα για την SEL Elections, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να συμμορφωθούν Τι θα γινόταν λοιπόν αν αυτοί πήγαν και πήραν τα δεδομένα μου από τους ε, ε, διακομιστές. Ε. Σε κάθε περίπτωση εγώ έχω μία απέτηση η οποία υποβλήθηκε στο Ανώτο Δικαστήριο βάσει του τμήματος 7 του DPA στις 16 Μαρτίου 2018 με την οποία γίνεται μία, υπάρχει ένα αίτημα να ανακτήσω τα δεδομένα μου. Κάτι αίτημα το οποίο έχει, δεν έχει ικανοποιηθεί. Ζητάμε λοιπόν να υποχρεώσει το δικαστήριο την SCL Elections ε, να αποκαλύψει στοιχεία για τους ψηφοφόρους και το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δικά μου ε, στοιχεία ώστε να αναγνωρίζομαι εγώ σε ένα σύνολο δεδομένων ώστε να συμμετιστεί ένα μοντέλο των πολιτικών μου πεπιθήσεων και των τάσεων. Παρότι πολλοί υπάλληλοι της Cambridge Analytica αναφέρουν ότι έχουν 5.000 σημεία δεδομένων αναψηφοφόρο και ψυχογραφικά προφίλ, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει τις απαιτήσει ε, βάσει του τμήματος 7 του DPA. Ε, λέγεται λοιπόν τα δεδομένα που ελήφθησαν σε αυτά τα αρχεία ε, ψηφοφόρων ήταν περαιτέρω των απλών, πέρα των απλών δημογραφικών ε, στοιχείων. Εδώ εμφανίζονται διάφορα νέα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ξέπλυμα δεδομένων όπου δεδομένα παράνομα ε, πέφτουν σε χέρια ε, πέραν των συνόρων και χρησιμοποιούνται ενδεχομένω για παράνομου σκοπού, όπου βρώμικα, για να το πούμε έτσι, δεδομένα να με καθαρά δεδομένα για να τα ξεκαθαρίσουν. Και είναι ένα νέο πρόβλημα αυτό που, η... που μας δείχνει η ιστορία αυτή της Cambridge Analytica, της GSR και του Facebook. Γι' αυτό έχει κλονίσει τον κόσμο. Παρότι είναι δύσκολο να εξηγήσουμε το γιατί, διότι σχεδόν όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ένα, ε, εδώ έχουμε ενδεχομένω ένα έγκλημα κατά της δημοκρατίας βάσει δεδομένων. Η προσωπική αυτονομία, η εθνική κυριαρχία πολιορκούνται αυτή τη στιγμή με όλους τους ε, νόμους που έχουμε ως ασπίδες και εγώ ως πολίτης ενός κράτους που δεν δίνει στους πολίτες τα απαραίτητα δικαιώματα για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας με, από τη νέα μικροστόχευση και τον ε, πόλεμο των πληροφοριών ε, που μένεται αυτή τη στιγμή. Εάν εγώ δεν μπορώ να τραβήξω τα δικά μου δεδομένα από όλο αυτό το συνονθήλευμα δεδομένων και δεν μπορούν να κάνουν και άλλοι, απομένουν πολλά να γίνουν για να προστατεύσουμε απόλυτα του ανθρώπου, ειδικότερα σε περίπτωση ε, εγκλημάτων βάσει δεδομένων. Όταν οι οργανισμοί προσπαθούν λοιπόν να ρίξουν αλλού την ευθύνη Εξακολουθώ να παρακολουθώ την υπόθεση της Cambridge Analytica. Πρόκειται για μια ιστορία αποφυγής ή ευθύνης. Δεν μπορώ να το καταλάβω τελικά. Έχουν διάφορα ε, δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους Αμερικανοί πολίτες χάρη στους Ευρωπαίους, χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όλα αυτά τα δεδομένα για τους ψηφοφόρους που περνούν μέσα από όλες αυτές τις βιομηχανίες ε, χειραγώγησης των εκλογών ε, του Facebook και ε, διαφόρων στρατιωτικών ε, οργανισμών που χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα. Η πρόσφατα αποκαλυφθήσα Sile Group που παρέχει πληροφορίες για διάφορους πελάτες ε, για κέρδος και απόκτηση δύναμης. Όλοι αυτοί παραβιάζουν την προστασία δεδομένων το ιδιωτικό απόρριτο είναι τα νέα αυτά ε, δεδο... Ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε εγκλήματα κατά μεγαλών πληθυσμών. Η μικροστόχευση, το micro-targeting χρησιμοποιείται για μικροεπιδράσεις την περασμένη εβδομάδα. Η συνάντηση, η συνέλευση ε, μετόχων του Facebook εκεί αναρωτήθηκαν κατά πόσο θα υπάρξει πρόβλημα σε επενδύσεις και κατά πόσο έχουν παραβιαστεί μαζικά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταστήσει σαφές ότι τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας ε, αντιλαμβάνονται ότι υφίστανται τη δικαιοδοσία, βρίσκονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των χωρών όπου δρούν. Χώρες λοιπόν με ανύπαρκτα ή πολύ αδύναμα καθεστώτα προστασίας δεδομένων ήταν βασική στόχη όπως οι ΗΠΑ σε τέτοιου μορφή παρέμβαση στις εκλογές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να αποτρέπονται όσοι θέλουν να αναμειχθούν στις εκλογές ε, και να αποφεύγονται οι παραβιάσεις ευρείας κλίμακας. Πόσο ο υπάρχον κανονισμός προστασίας δεδομένων βοήθησαν να ε, προστατευθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ξένες επιδράσεις και από τις ε, ψευδείς εκλογικές εκστρατείες. Πώς τα εργαλεία που χρησιμοποίησε το Facebook για τους διαφημιστές και για τις πολιτικές εκστρατείες όπως το Custom Audiences και το Lookalikes χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα όχι μόνο από ξένες δυνάμεις αλλά και από φαινομενικά ε, θεμητούς ε, ε, παράγοντες εκλογικών εκστρατιών και άλλων. Ελπίζω να σας ενημέρωσα επαρκώς για τους πιθανώς μη αναμενόμενους δικαιούχους του μοντέλου ε, αυτού προστασία δεδομένων της Ευρώπης. Ελπίζουμε να μεγαλώσει η επίδρασή του μετά το GDPR. Η ιστορία μου είναι ένα μόνο παράδειγμα για το πώς ε, ένας τυπικός Αμερικάνος ε, ε, βρίσκεται πιο εκτεθειμένο στην Αμερική σε σχέση με την Ευρώπη όπου υπάρχουν ρυθμιστές με τα απαραίτητα εργαλεία, με ποινικέ δυνατότητες, με δυνατότητες κατάσχεσης ώστε να αποτραπούν μελλοντικοί κακόβουλοι παράγοντες από το να προσπαθήσουν με λογισμικό διεισδυτικό να συνδυάσουν δεδομένα, να χειραγωγήσουν εκλογικά σώματα με τα εργαλεία του μάρκετινγκ, με στρατιωτικές μεθόδους ώστε να επιλέγουν κινητοποίηση ή αποκινητοποίηση εκλογέων. Η μικροστόχευση θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την επιρροή των εκλογικών σωμάτων αλλά αυτές οι μηχανές πολιτικής τεχνολογίας βασίζονται στα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, στην προστασία, στην πρόσβαση ε, βάσει του σχεδιασμού τους. Η τεχνολογία θα πρέπει να προχωρήσει, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει από την καταστροφή της Cambridge Analytica. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Και τέλος ο Κρίστοφερ Βάιλι που μας αποκάλυψε την υπόθεση και πρώην Διευθυντής Ερευνών της Cambridge Analytica. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριες ε, και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω μαζί σήμερα. Είναι η πέμπτη μου κατάθεση σε νομοθετικό σώμα και ίσως η πιο σημαντική. Ο κόσμος δρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, όπως είχε και ο Ζαν Μονέ, και αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη μόνο σε κατάσταση κρίσης. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι υπάρχει κρίση. Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο κρίση ιδιωτικότητας, αλλά ίσως οδήγησε στην, στο να χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της. Αυτό το οποίο είδα εγώ στην Cambridge αναλυτικά πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Η Cambridge Analytica είναι το πρώτο αυτό σημάδι του νέου ψυχρού πολέμου που εμφανίζεται. Ήμουν διευθυντή ερευνών ε, από το 2014 μέχρι το 2018. Η SEL Group είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει στρατιωτικά έργα και η Cambridge Analytica ιδρύθηκε με λεφτά του Ρόμπερτ Mercer ε, ο οποίος εγκατέστησε τον Steve Bannon ως αντιπρόεδρο με ευθύνη να διχειρίζεται την εταιρεία στις καθημερινές τη λειτουργίες, αλλά δεν τον απασχολούσε μόνο η, η Αμερική. Ο κ. Μπάνον ε, είδε και τη Μεγάλη Βρετανία ως ένα βασικό σημείο. Το ήθος τη εταιρεία ήταν ότι όλα επιτρέπονται. Είδα προσωπικό της εταιρεία να προσπαθεί να αποσπάσει λεφτά τα οποία πήγαιναν προς μια αφρικανική χώρα προς όφελος συγκεκριμένου πολιτικού. Η εταιρεία λοιπόν οδηγούσε σε διαφθορά και ένα, μια απεικιοκρατία του 21ου αιώνα. Μεταξύ του 2013 και 2015 η Cambridge Analytica χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα που λεγόταν Project Ripon που στόχο είχε να αναπτύξει αλγόριθμους ψυχολογικών προφίλ για πολιτικές εκστρατείες. Για να είμαστε σαφείς, η δουλειά του, της Cambridge Analytica δεν είναι παραδοσιακό marketing όπως λένε κάποιοι είναι λανθασμένη η ισοδυναμία αυτή και παραπλανητική. Η Cambridge αναλυτικά ειδικευόταν στην προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Έβρισκαν νοητικές και ψυχολογικές αδυναμίες τις οποίες εκμεταλλεύονταν μέσω κάποιων πληροφοριών όπως παραδείγματο χάρη τις νευρώσεις, την παράνοια και τις ε, προκαταλήψεις. Για όσους λένε ότι δεν λειτουργούν τα προφίλ, έχουμε πάρα πολλές έρευνες ε, σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, όπως το Proceedings of the National Academy of Sciences ε, και άλλα. Ακόμα και το ίδιο το Facebook έχει μία ένα δίπλωμα έβρεση τεχνίας ε, το οποίο αφορά όπως λέει χαρακτηριστικά την διαμόρφωση ψυχολογικών προλήγων. Ο Dr. Alexander Κόγκαν ήταν αυτός ο οποίος ανέπτυξε τις μεθόδους μας ε, και τις σχετικές ε, εφαρμογές ε, που συνέλεγαν δεδομένα του χρήστη και των φίλων του χωρίς την συγκεκριμένη τους συνένεση, κάτι το οποίο επέτρεπε το Facebook τότε. Αργότερα έμαθα μέσω της επικοινωνίας με το Facebook πως δεν είχε την ανάλογη άδεια ο κύριος Κόγκαν για εμπορικές ή πολιτικές δραστηριότητες. Όμως οι όροι χρήσης της οδηγίας έλεγαν ότι τα δεδομένα αυτά θα απολυθούν σε τρίτα μέρη και το Facebook αντέγραψε μάλιστα και είχε και αντίγραφο αυτών των όρων χρήσης τους οποίους ενέκρινε και επέτρεψε στην εφαρμογή να συλλέγει αυτά τα δεδομένα με αυτούς τους όρους χρήσης. Όταν ερωτήθηκε το Facebook, ο τεχνικός διευθυντής ε, του Facebook παραδέχτηκε ότι δεν διάβαζε όλους τους ε, όρους χρήσης. Μια εταιρεία μάλιστα η οποία περιμένει οι χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης ενώ δεν το κάνει το ίδιο το Facebook. Εάν είχαν διαβάσει τους όρους του Δόκτωρα Κόγκαν ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η SCL Group κατόπιν ε, συνέστησε μια εταιρεία ονόματι Aggregate IQ, η οποία έφτιαξε την πλατφόρμα που συνέλεγε τα δεδομένα του Facebook. Πρώτα από όλα. Έγινε μια δοκιμή στο Trinidad εκεί πέρα. Στόχο είχε να συλλέξει δεδομένα για να παρακολουθεί τις συνήθειες ε, σερφαρίσματος στο διαδίκτυο των Χριστών στην Καραϊβική. Επίσης ε, αναζήτησε άνωνυμα τα δεδομένα των Χριστών το 2015 επίσης ελήφθησαν κάποια βίντεο, βίντεο με συγχωρείτε, τα οποία έδειχναν κάποιες δολοφονίες και ακροτηριασμούς ψηφοφόρων, τα οποία φρόντισε να εξαφανίσει. Το 2016 η ίδια εταιρεία έλαβε το 40% της χρηματοδότησης του Vote Leave. Τα περισσότερα από αυτά πήγαν σε στοχευμένες διαφημίσεις μέσω Facebook και από άλλε εκστρατείε, όπως το DUP, το Believe και του Βετεράνου για την Βρετανία. Και το DUP μάλιστα δόρισε και 625.000 λίρες για να χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες της Και Υπάρχουν συγκεκριμένα και αυστηρά όρια εξόδων στην Βρετανία και απαγορεύεται ο συντονισμό των εκλογικών εκστρατιών. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ακριβώ συνέβη στο δημοψήφισμα. Το Vote Leave έστησε νέες ε, εταιρείε και εκστρατείε και τους δόρισε λεφτά με αποτέλεσμα να παραβιάζει τα όρια της χρηματοδότησης. Το Facebook έχει επιβεβαιώσει στην έρευνα του Βρετανικού Κοινοβουλίου πως το AIQ δημιουργούσε παρόμοια προφίλ ε, για τις διάφορες εκστρατείες. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια έρευνα εν εξελίξη για παράνομες δαπάνες και για εγκλήματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα. το ανακοινώθηκε πέρσι ότι γινόταν η έρευνα, το Vote Leave μπήκε σε έναν σκληρό δίσκο του Believe. Και όταν δημοσίευσε την υπόθεση ο Guardian τον Μάρτιο, υπήρξε πάλι πρόσβαση στον ίδιο κοινόχρηστο δίσκο. Και φαίνεται ότι προσπαθούσαν να παραποιήσουν τα δεδομένα. Εμπλέκεται εδώ και το γραφείο της Πρωθυπουργού. Δύο σύμβουλοι της Τερέζα Μέη είχαν εργαστεί στην ε, υπόθεση χρηματοδότησης της AIQ, ξέρουν λοιπόν τι συνέβη και προσπαθούν να καθυστερήσουν την έρευνα μέχρι να οριστικοποιηθεί το Brexit. Επρόκειτο λοιπόν για την μεγαλύτερη δαπάνη του vote leave. Δεν πρόκειται για κάτι το μικρό. Φαίνεται ότι ακριβώς προσπάθησαν να παρακάμψουν τον εκλογικό νόμο. Η Cambridge Analytica διαλύθηκε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της θα αισθάνονται τον αντίκτυπο για πολλά χρόνια. Θεωρώ πως δεν θα είχε συμβεί το Brexit εάν δεν τα είχε κάνει αυτά η Cambridge Analytica. Επίσης ε, δεν θεωρώ ότι το αποτέλεσμα του Brexit ήταν κάτι το οποίο έγινε δίκαια. Και περίεργως το Βρετανικό δίκαιο δεν προσφέρει κάποια δυνατότητα επανόρθωσης. Αν επρόκειτο για κάποια βουλευτική έδρα θα γινόταν επανάληψη της εκλογής. Αλλά για δημοψήφισμα αυτό δεν προβλέπεται γιατί κανείς δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπήρξε συστηματική εκλογική απάτη και από ξένες εταιρείε και όσον αφορά την χρηματοδότηση. Αυτό το επέτρεψε το Facebook και ο Μάρκ Ζαγκερμπέργκ αρνείται να απαντήσει κάποιες κέρυες ερωτήσεις για τα όσα συνέβησαν στο Brexit. Αν γινόταν αυτό στην Ιγυρία ή στην Ζιμπάμπουε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτούσε επανάληψη της ψηφοφορίας. Ίσως πρέπει να ζητήσουμε το ίδιο και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο 2 της ε, συνθήκης του Μάστριχ λέει πως ε, οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ λέει ότι όπου υπάρχουν εκλογές πρέπει να είναι ελεύθερες και δίκαιες. Το Brexit δεν είναι εσωτερικό ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συμμορφώνεται στι δημοκρατικέ απαιτήσει Ένωση. Έχει λοιπόν δικαίωμα και υποχρέωση να γνωρίζει εάν εκατομμύρια Βρετανοί πολίτε θα σταματήσουν να είναι Ευρωπαίοι πολίτε λόγω κάποια εκλογική απάτη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να μείνει ή να φύγει, είναι ένα ζήτημα κράτου δικαίου και στη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί μια μεγάλη συνταγματική αλλαγή, τη μεγαλύτερη εδώ και μια γενιά. Και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει ένα μέλος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα πάντα έχουν γίνει σωστά και χωρίς αμφισβητήσεις. Στο Facebook βεβαίως για πρώτη φορά ειδοποιήθηκε το 2015 για την Cambridge Analytica. Δεν προειδοποίησε τότε τους ε, χρήστες και ανέλαβε βεβαίω δράση μόνο α, τρεις εβδομάδες αφότου ο Guardian έγραψε για την ιστορία. Και η αντίδρασή του ήταν να μηνύσει την Guardian, προσπάθησαν να εκφοβήσουν και εμένα και να μην δημοσιοποιηθεί η ιστορία την οποία ήξερε βεβαίω ότι ισχύει. Ο τεχνικός διευθυντής του Facebook προσφάτως στην έρευνα δήλωσε ότι η εταιρεία είχε υποθέσει ότι η απειλή δημοσιογράφων είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απογοητεύτηκα από το πώς έδρασε το Facebook πριν δημοσιοποιηθεί η ιστορία. Προσφέρθηκα να βοηθήσω και είπε ένας αντιπρόεδρος τους, στους δικηγόρους μου, ότι βεβαίως ήταν υπέρ της συνεργασίας. Τελευταία στιγμή όμως ε, έβγαλα μια εκείνωση τύπου ότι με είχαν αποκλείσει από την πλατφόρμα. Παρέμενα αποκλεισμένος από το Facebook παρά το ότι επέμενε ο επόπτης προσωπικών δεδομένων ότι δεν ήμουν αντικείμενο έρευνας. Και απαντώντας εξ ονόματος της Βρετανικής κυβέρνησης, ε, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι είναι κάτι το εξωφρενικό. Αυτό δείχνει ακριβώς την απεριόριστη ισχύ που έχουν οι πλατφόρμες έναντι των χρηστών, όταν κάποιος μπορεί πολύ απλά να διαγραφεί. Δεν υπάρχει κάποια σωστή διαδικασία, δεν υπάρχει έλεγχος της πλατφόρμας. Και τι γίνεται στην δημοκρατία όταν κάποιοι οι οποίοι τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους απλά διαγράφονται. Το Facebook λοιπόν δείχνει και τις τεράστιες ε, συνέπειες του ότι σιγά σιγά υπάρχει μια συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην Silicon Valley. Παραδείγματος χάρη διαγράφηκε και ο λογαριασμό μου από το Instagram παρά το ότι δεν είχε καμία σχέση. Απλά κοινή ιδιοκτησία πλέον ανοίξει στο Facebook. Το Facebook απέτησε να δώσω τον προσωπικό μου υπολογιστή και τηλέφωνο. Η εταιρεία αγνόησε το ότι είχα δώσει ήδη στοιχεία στις αρμόδιες Βρετανικές αρχές. Στην ουσία το Facebook απαιτούσε να τους δώσω τα στοιχεία τα οποία ήταν αντικείμενο της έρευνας. Δεν τους ενδιέφερε η ορθή δικαστική διαδικασία των αρμοδίων αρχών. Επίσης, στο Facebook αγνόησε το ότι χρειαζόμουν πρόσβαση στον λογαριασμό μου για να δώσω στοιχεία στις Βρετανικές αρχές. Για να δώσω στοιχεία παραδείγματο χάρη στην έρευνα τη εκλογική επιτροπή. Και όλα αυτά επειδή δεν είχα πρόσβαση στον λογαριασμό μου στο Facebook. Δεν του ενδιέφερε ότι εμπόδιζαν την έρευνα. Αλλά όπω είδαμε, με την συνεχόμενη άρνηση του Μαρκ να έρθει να καταθέσει στην Βρετανία, είναι αδύνατον οι χώρες να κάνουν αυτές τις εταιρείε να λογοδοτήσουν. Και τώρα το η Βρετανικό Κοινοβούλιο εξετάζει την πιθανότητα να εκδώσει μια διαταγή προσαγωγής του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική νοοτροπία. Η τεχνολογία πρέπει να επιβλέπεται δημοσίω. Δεν μπορεί να απαλλάσσεται από αυτό επειδή είναι λογισμικό κάθε χρόνο. Αγοράζουν οι Ευρωπαίοι περισσότερε συσκευέ που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Σύντομα, το διαδίκτυο των πραγμάτων θα είναι φυσιολογικό στα σπίτια μα. Αλγόριθμοι θα οδηγούν τα αυτοκινητά μα, θα οργανώνουν τι ζωέ μα. Το GDPR είναι μια καλή απόπειρα δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά εξακολουθεί να έχει πολλέ αδυναμίες. Το GDPR απαιτεί ιδιωτικό απόρριτο από σχεδιασμό, αλλά τι γίνεται με τη διαφάνεια. Δεν ξέρουμε τι διαφημίσει θα στέλνονται σε συγκεκριμένους χρήστες ε, ε, μέσων κοινωνική δικτύωσης. Ε, αν αυτό χαρακτηριζόταν από διαφάνεια θα μπορούσε να το ελέγξει ο καθένα. Τα διασυνδεδεμένα συστήματα επίση δημιουργούν πρόβλημα ε, αυτό θα χαρακτηρίζει το μέλλον ε, της όλο και μεγαλύτερης διασύνδεσης. Πώς θα ελέγχει κανείς ένα σύστημα όταν υπάρχει ε, σύνδεση μεταξύ όλων των συσκευών μεταξύ τους. Τι γίνεται με τα δεδομένα σε δυναμικά δίκτυα όπου υπάρχουν τόσοι μετασχηματισμοί, προσκλήσεις, ανταλλαγές δεδομένων. Ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. αν θέλετε να, κάνετε να πείτε ένα συμπέρασμα... okay, I know, I'm the villain and you. That's fine. Um... You get a... Ναι, ναι, αν κατακλείδη να πω ότι <laughs> έχουμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και ξεκινάνε όλα από εσά. <laughs> I'm just about to really... Πρόεδρος. Εγώ τώρα θα μιλήσω για αυστηρά όρια ε, για το χρόνο μιλία των Ευρωβουλευτών. Ένα λεπτό για την ερώτηση και σας παρακαλώ, πολύ δυσκολευθήκαμε για να το καταφέρουμε αυτόν τον κατάλογο. Παρακαλώ να μην το αφισβητήσετε, είναι ένας κατάλογος και είναι δίκαιος από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό για την ερώτηση και όταν την υποβάλλετε θα πρέπει να διευκρινίσετε σε ποιον την υποβάλλετε την ερώτηση. Ποιος θέλετε να την απαντήσει και για την απάντηση θα έχετε δύο λεπτά. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε και να μην ε, επικριθούμε για το τι έγινε και την άλλη φορά. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επιτροπές. Έχουμε πρώτα την Μπάρμπαρα Σπινέλη για την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Αντιπροσωπεύει τον Πρόεδρο της ΑΦΚΟ. Εγώ επιβάλλω μια ερώτηση εξ ονόματος της κυρίας Χούμπνερ, που είναι ε, η πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Και η ερώτησή μου απευθύνεται στην κυρία Ελίζαμπεθ Ντένον σε αυτή την ψηφιοποιημένη εποχή πώς μπορούμε εμείς ως νομοθέτες να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη χρήση της, των ευκαιριών που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες για να συνδέονται και να ενημερώνονται ανοιχτά οι εκλογές για τις επιλογές τους και τους κινδύνους που μπορεί να ενυπάρχουν και να, δηλαδή να επηρεαστούν από αδιαφανείς και πιθανά παράνομους τρόπους. Ευχαριστώ. Κυρία Ντένα, με δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στην έκθεση επί της οποίας εργαζόμαστε και που θα ανακοινωθεί αργότερα το, αυτόν μήνα αυτό, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αξία των κοινωνικών μέσων και της επιγραμμικής επικοινωνίας για τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα που έτσι μπορούν να συνδεθούν με τους ψηφοφόρους και να ενθαρρύνουν τη δημοκρατική συμμετοχή. Ταυτόχρονα αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο και διαφανή τρόπο και επίσης πρέπει να γίνει με νόμιμο τρόπο. Όταν ε, εμείς ε, ε, πήραμε, ε, συνομιλήσαμε με όλα τα κύρια πολιτικά κόμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τους μιλήσουμε, για να δούμε πώς χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα και πώς αναλύουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να στοχεύσουν σε ομάδες ανθρώπων. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει πολλά πράγματα και το τι ακριβώς συμβαίνει ε, επί τόπου. Μας είπαν επίσης ότι πιστεύουν πως η τεχνολογία έχει ξεπεράσει τα θέματα της ιδιωτικής ζωής, της διαφάνειας και της ηθικής σε το χώρο. Οπότε ε, ε, είναι καιρός να δούμε την αθήκη πλευρά, να δούμε τη διαδικασία, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων για μικροστόχευση των ατόμων. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να μας ακολουθήσει, να μην δημιουργήσουμε δηλαδή κάποια χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει πραγματικά δημόσια συζήτηση για κάποιο ζήτημα. Φτιάχνουμε λοιπόν μια έκθεση για έναν κώδικα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, κώδικα διοντολογίας για τις πολιτικές εκστρατείες, για τα πολιτικά κόμματα, για τη χρήση των δεδομένων και τις ανάλυσης δεδομένων. Και νομίζω πως πολλές θετικές, ε, ε, θετικά σχόλια λαμβάνουμε από τους πολιτικούς και τα πολιτικό κόμματα για τις λεπτομέρειες που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. κυρία Λάουρα Φεράρα. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι προ τον κύριο Κρίστοφερ Βάιλι. Έτσι θα μπορέσετε να συνεχίσετε και την ομιλία σα, Η πρόσφατη εξέλιξη τη τεχνητή νοημοσύνη θέτει διάφορα ε, νομικά και ηθικά ζητήματα για του χρήστε. Ε, ε, πολλά περιεχόμενα λαμβάνονται και αναλύονται. Μπορείτε να διευκρινίσετε πώ πραγματοποιήθηκε αυτή η ανάλυση στην πρακτική. Έγινε κάποια συζήτηση περί νομιμότητας και ηθικής σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Κρίστοφερ Βάλι για δύο λεπτά. Για να καταλάβω αυτό που ρωτήσατε, εννοείται πώς έγινε και αν ελήφθησαν υπόψη ε, οι χρήστες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πολλά δεδομένα αποκτήθηκαν ε, μέσω του συστήματος του Facebook στο οποίο αναφέρθηκα, αλλά και μέσω προμηθευτών του Facebook και διαμεσολαβήτρες εταιρείε. Όλες αυτές οι πληροφορίες ε, συγκεντρώνονται σε ένα μητρό βάση δεδομένων για να δημιουργήσει μια εικόνα των πολιτών. Βλέπει κανείς δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι online, σε τι δαπανούν χρήματα που ζουν, αν έχουν ε, πάρει κάποιο ε, δάνειο για παράδειγμα αγορά τα κτλ. Και με βασικές πληροφορίες όταν κάποιος απαντά σε κάποιες ψυχολογικές έρευνες εκεί ψάχνει να βρει κανείς ε, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων. Έτσι ε, έχουν σχεδιαστεί αυτοί οι αλγόριθμοι και σχετίζονται αυτοί μετά με την πλατφόρμα στόχευσης του Facebook για να στοχεύσουν συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ πολλές φορές έχω θέσει το ζήτημα της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Θεωρήθηκα ότι δεν ελειφθεί υπόψη, πολύ ειλικρινά. Ε, εγώ από πλευρά μου ήθελα να τεθεί αυτό το θέμα τη συμμόρφωση ε, με του κανονισμού προστασία δεδομένων, όχι μόνο όσον αφορά του Ευρωπαίου πολίτε, αλλά με οποιονδήποτε βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και που για κάποιο λόγο έχει τα δικαιώματα αυτά. Ωστόσο, αγνοήθηκα, δυστυχώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σον Κέλλη, πρόεδρος, εκπροσωπεί τον πρόεδρο τη Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές. Ε, πολύ ενημερωτική. Ένα σχολείο πρώτα απ' όλα. Έχουμε έναν πρώην υπαλλό του Facebook και της Cambridge Analytica εδώ. Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Επίσης ε, συζητήθηκε εσωτερικός έλεγχος για την εξέταση των παραβιάσεων των δεδομένων, ναι, δεν θα μπορέσει να υπάρξει εξωτερικό ε, απαραίτητα έλεγχο και μετά ο Μάρκ Τζούκερμπεργκ. Εγώ επειδή έχω εργαστεί ως συζητητής για το GDPR και πήγα και στη Silicon Valley πριν από δύο εβδομάδες, άκουσα επένους για τον GDPR, μα είπαν ότι θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο ο κανονισμός αυτός και ταυτόχρονα ακούμε ότι οι χρήστες από την Αυστραλία, την Αφρική, την Ασία δεν ε, εντάσσονται στον κανονισμό. Τι έχετε να πείτε για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, κύριος Παρακλάς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που αφορά τον έλεγχο των εφαρμογών ή κάποιων εφαρμογών που ενδεχομένως έχουν παραβιάσει τους όρους του Facebook, συμφωνώ με αυτό που λέτε, είναι προτιμότερο να γίνει με εξωτερικό έλεγχο. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχουμε στον τομέα της τεχνολογίας είναι η έλλειψη διαφάνειας, όχι μόνο για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, αλλά και για τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Συμφωνώ λοιπόν, ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγματοποιείται εξωτερικά από κάποιον που δεν αμείβεται από το Facebook. Τώρα όσον αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση. Δεν είμαι βέβαιος ότι Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ουσία της ερώτησης. Τι ακριβώς ε, προσπαθείτε να καταλάβετε. Ακούγεται ότι πρέπει να περιορίσει, θέλει να περιορίσει τη χρήση του GDPR το Facebook, ε, αποκλείοντας κάποιους χρήστες ε, σε άλλες υπήρους που παλιότερα χρησιμοποιούσαν όρου οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί στην ε, Ιρλανδία. Συγγνώμη δηλαδή, η ερώτησή σας είναι κατά πόσο αυτό θα πρέπει να επιτραπεί στο πλαίσιο του GDPR ή γιατί το κάνει αυτό η εταιρεία. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να, μπούμε, να ξεκινήσουμε διάλογο, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, επειδή το GDPR ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει κάποια αντίφαση. Δηλαδή, ε, αφενό ε, επενούν το GDPR και λένε πρέπει να εφαρμοστεί παγκοσμίω και μετά αποκλείουν όλου αυτού του λαού που ε, ενώ ίσχυε για αυτού το καθεστώ τη Ιρλανδία, του λένε ότι ισχύει το καθεστώ εκτό Ευρώπη τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πράγματι λέει ο κ. Παρακελάς. Δεν είναι στο πνεύμα του GDPR, ούτε στο πνεύμα αυτού που περιγράφουν αυτοί να εφαρμόσουν δηλαδή, να εφαρμόσουν δηλαδή παγκοσμίω τι προστασίε που προσφέρει το GDPR. Σε περίπτωση που ήθελα πραγματικά να δράσουν με αυτό το πνεύμα, δεν θα είχαν μετακινήσει τους λογαριασμούς αυτούς. Εκρεμεί και ένα άλλο ερώτημα. Πώς καθορίζει κανείς τα δεδομένα σε ένα μήνυμα μεταξύ ενός Ευρωπαίου πολίτη και ενός πολίτη που δεν είναι Ευρωπαίος. Πού ανήκουν αυτά τα δεδομένα, σε ποιο καθεστώς εντάσσονται. Όλες αυτές οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα επιληθούν ε, στις ε, δίκες, ε, στις δικαστικές διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Σας έδωσα λίγο παραπάνω χρόνο γιατί χρειάζονταν αυτές οι εξηγήσεις. Επόμενη ερώτηση από τον πρόεδρο Λίμπε. Ε, εγώ αυτό αυτοπροσώπως είμαι μόνος πρόεδρος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω την ερώτησή μου προς τον κύριο Κρίστοφερ Βάιλι. Ωραία. Λοιπόν, δεδομένων των όσων ξέρουμε και των όσων είπατε, Κρίστοφερ, για τον αντίκτυπο της ε, Brexit, αναλυτικά μιλήσατε για το δημοψήφισμα του Brexit και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις αναφέρατε την εταιρεία MR Data που συνέστησαν πολλά άτομα που συμμετείχαν και στην Cambridge Analytica και τη μητρική εταιρεία την SCL Group. Υπάρχουν πολλά ίδια άτομα και σε αυτή την εταιρεία. Ποια είναι η πιθανότητα, θεωρείτε, περαιτέρω χρήσης αυτών των αλγορίθμων που επηρέασαν τις εκλογές ε, μέσω του προφίλ μεμονωμένων ψηφοφόρων. Βλέπετε να επαναλαμβάνεται αυτό και σε άλλες εκλογές, γιατί βεβαίως έχουμε και ένα ακροατήριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μάλιστα είναι διπλή ερώτηση από ό,τι βλέπω, δηλαδή τι θα γίνει με τους αλγοριθμούς και δεύτερον τι έχει κάνει η εταιρεία σε άλλες χώρες, κατάλαβα καλά, μάλιστα. Είμαι επιφυλακτικός ε, για το εάν η εταιρεία πραγματικά θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, αλλάζει μεν ο Μανολιός, αλλά είναι ύποπτα, είναι ύποπτα το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν συστήσει και άλλες εταιρείε. Αν σκεφτούμε ότι έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να αναπτυχθούν αυτοί οι αλγόριθμοι και τα σετ δεδομένων, υπάρχει και οικονομικό κίνητρο να αποδώσει αυτή η επένδυση σε κάποια άλλη μορφή. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εικασίες βεβαίω για το τι κάνουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν είμαι πια εκεί. Όσον αφορά άλλες χώρες, ξέρετε, η εταιρεία πηγαίνει ανά τον κόσμο και κατά την άποψή μου έχει διαφύρει ευπαθείς δημοκρατίες για να εκμεταλλευτεί ευπάθειες ε, σε αυτά τα συστήματα ε, με σκοπό το κέρδος. Όμως κάποιες χώρες όπως ε, το Trinidad παίρνουν πολύ σοβαρά την υπόθεση και εξετάζουν το ότι μιλάμε για μια νέα μορφή απεικιοκρατίας μέσω των δεδομένων όπου μια χώρα μπλέκει στα εσωτερικά μιας άλλης. Απαντάει αυτό την ερώτησή σας. Ναι, πρέπει να απαντήσει γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, για την Επιτροπή ΙΜΚΟ η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Για ένα λεπτό ευχαριστώ Κλοντ και σας ευχαριστώ για αυτές τις ανατριχιαστικές ε, περιγραφές ε, του πώς κινδυνεύουν οι δημοκρατίες και οι εκλογικές διαδικασίες ε, και τα δημοψηφίσματα. Ακούσαμε πολλές συγγνώμε από το facebook ότι κάναν λάθος, δεν ήταν προσεκτικοί και θεωρούμε πραγματικά ότι η εμπορική ισχύς ε, πρέπει να πηγαίνει χέρι με χέρι με την ανάλογη ευθύνη. Αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει πέρα από τις παραβιάσεις δικαιωμάτων να δούμε και το θέμα αφαίρεσης του παράνομου ε, περιεχομένου. Λοιπόν, η ερώτησή μου απευθύνεται στην Ελίζαμπεθ τα μέτρα που λαμβάνει το Facebook ε, για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοια παραβίαση των δεδομένων επαρκούν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Ακούσαμε κάποιε πράξει. Ε, θεωρείτε ότι επαρκούν. Δεύτερον, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, εάν ληφθούν, από τα θεσμικά όργανα τη Ένωση ε, για να αυξηθεί η διαφάνεια. Και τρίτη ερώτηση, Πώ μπορούν οι πλατφόρμες να προστατεύσουν τα παιδιά μετά την χαμένη ευκαιρία του GDPR αυτού γιατί το Facebook ε, δημιουργεί προφίλ και παιδιών και τίθεται το ζήτημα βέβαια πιστοποίησης και της ηλικίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερώτησή σας για το εάν τα μέτρα που ανακοίνωσε το Facebook ε, για να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων επαρκούν, η απάντηση είναι ο καιρός θα δείξει. Υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει η έκθεσή μας ε, και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν νομίζω θα αποσαφηνίσουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο το Facebook αυτό το οποίο πρέπει να είναι πιο διαφανές και να συμμορφωθεί με την νομοθεσία, αλλά και άλλες πλατφόρμες ε, του διαδικτύου. Αλλά ο χρόνος θα δείξει για το Facebook. Ε, λοιπόν και πάλι υπάρχουν πολλές έρευνες που διεξάγονται μεταξύ των ομολόγων μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εποπτών Προστασίας Δεδομένων έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας. Η δεύτερη ερώτησή σας ήταν ποια μέτρα μπορούν να λάβουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων νομίζω είναι ένα σημαντικό πρωτοβήμα. Επίσης, τίθενται και ζητήματα δεοντολογίας που πρέπει να εξετάσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και γνωρίζω πως είναι εδώ πέρα και ο συνάδελφος, ο Τζοβάνι Μπερτορέλη, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το ζήτημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργεί ένα νέο κέντρο για την δεοντολογία των δεδομένων, γιατί αυτά τα ζητήματα δεν είναι πάντα άσπρα μαύρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα δεοντολογίας και γκρίζε ζώνες που πρέπει να εξετάσουν τα θεσμικά όργανα και οι βουλευτές. Η τελευταία σας ερώτηση, ο χρόνος, ναι, για τα παιδιά στο διαδίκτυο. Όπως ξέρετε, ο Γενικός Κανονισμός έχει ειδικού κανόνες για τα παιδιά που οι πάροχοι διαδικτύου πρέπει να σέβονται, δηλαδή θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών. Είναι ενδιαφέρον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, προβλέπει ότι η υπηρεσία μου θα πρέπει να αναπτύξει ένα κώδικα συμπεριφοράς για την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά. Μάλιστα, για την Επιτροπή Πολιτισμού, η πρόεδρος η Ζαμπίνε Φερχάιεν. Ναι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες ε, που λάβαμε και για τις απαντήσεις ε, Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, εκπροσωπώντας την Επιτροπή Πολιτισμού. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 10 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, την προστασία δηλαδή της επικοινωνίας των ΜΜΕ, έτσι ώστε παρά την χρήση ε, της ανάλυσης των δεδομένων που γίνεται με τρόπο σύνομο όταν δίνει την συνένεση του χρήστη να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων στην διάθεση του χρήστη. Πώς μπορούμε δηλαδή να εμποδίσουμε το να δημιουργηθούν ε, κάποιοι διάβλοι μονομερείς, ε, όπως είδαμε στην περίπτωση, μονομερούς ενημέρωσης δηλαδή, όπως είδαμε στην περίπτωση του Brexit και άλλων εκλογών που είχαν μεγάλη επιρροή. Δεν απευθυνθήκατε σε κάποιον ε, να απαντήσει, Κάρολ. Δεν είμαι σίγουρη ε, αν απευθύνεται στον ε, κύριο Παρακύλας ή στον κύριο Γουάιλι. Απαντήσω κύριο Παρακύλας. Να προσπαθήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ ότι η μονομερής ενημέρωση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι οι εταιρείε οι τεχνολογικές πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό. Ε, για να είμαι σαφής, μιλάω για το ότι περιβάλλονται οι χρήστες με απόψεις με τις οποίες ήδη συμφωνούν μόνο. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Ένα δεύτερο μέρος του προβλήματος είναι ότι όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, όταν φτιάχνουμε αλγόριθμους που καταλήγουν σε κάτι τέτοιο. Επίσης μπορούν ε, να διαδοθούν ε, σε ειδήσει, ε, θεωρίες, συνωμοσίες κλπ. Οπότε έχουμε αφενός την πλευρά των εταιρείων τεχνολογίας που ιστορικά δεν ασχολήθηκαν με αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι τώρα το κοιτάνε πιο πολύ βάθος, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να κάνουν. Και υπάρχει και η πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στο πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και τι αποτέλεσμα έχουν. Δηλαδή να απαιτούμε από τις εταιρείες να μας δίνουν στοιχεία για το τι μορφή έχει το πρόβλημα και αυτό από μόνο ότι είναι μια αρχή για να λυθεί. Σας ευχαριστώ η Ρομπέρτα Μετσόλα για την ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα δεδομένα πλέον είναι ο χρυσός ε, της εποχής μας ε, και βλέπουμε ότι ασυνείδητοι, οι πολιτικοί και όσους τους στηρίζουν ε, θα τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προπαγάνδα και να κάνουν την προπαγάνδα να φαίνεται ως γεγονός. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι παραθυράκια υπάρχουν ακόμα. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν αφορά μόνο την κατάχρηση δεδομένων, αλλά για ένα σύστημα το οποίο και συστήματα τα οποία οικοδομήθηκαν για καλό και χρησιμοποιούνται εναντίον μας. Ε, εγώ με Μαλτέζα και εκεί είχε κάποιον ρόλο η Cambridge Analytica, ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα δεδομένα 6.000 Μαλτέζων πολιτών και εκατομμυρίων Ευρωπαίων και ποιος ε, ζήτησε κάτι τέτοιο. Ε, το ερώτημά μου απευθύνει στην κυρία Καντουόλτα. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε από εδώ ε, τους δημοσιογράφους ε, και τους καταγγέλλοντες και με κατόπιν στον κύριο Παρακύλες. Τι, αυτό, μία ερώτηση έχω. Μα μάλιστα, εντάξει, καλώς. Να προσθέσω λοιπόν, αν α, ε, μπορεί. Ρομπέρτα τώρα, αφού ξέρεις. Λοιπόν, ναι, τι μπορώ να κάνω για να επαναληφθεί ξανά αυτό το φαινόμενο. Μα με, με κοίταγες τώρα, αφού ξέρεις. Λοιπόν, Κάρολ για δύο λεπτά. Όπως είπα και στην εισήγησή μου, πιστεύω πως είναι τόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Ε, δείχνει ε, απελπισία από το Facebook το να μιλά μόνο για το μέλλον και να προχωράει. Πάντως εγώ πιστεύω πως αν δεν καταλάβουμε απολύτως τι ακριβώς συνέβη σε αυτές τις πολύ κρίσιμες εκλογές και ακριβώς πώς η εκλογική μας νομοθεσία δυνητικά παρεκτρά, μάλλον ε, παραβιάστηκε, ε, δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά και φυσικά και αυτό επηρεάζει το δικό σας μέλλον και το μέλλον όλων μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ρίξετε έναν προβολέα σε αυτή την υπόθεση Όλες αυτές οι έρευνες που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολλές, πολλές έρευνες από πολλές αρχές. Όλες συνδέονται και όλες έχουν κοινό σημείο την Cambridge Analytica και όλες τις ε, συνδεδεμένες με αυτήν ε, εταιρείε. Και όλες συνδέονται με τον Robert Mercer και τον Steve Bannon, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Και με τον Νάιτζελ Φαράζ ε, που σίγουρα εκείνος έχει ε, πολλά στοιχεία και μπορεί να φωτίσει αυτή. Δεν απαντάει όμως στους δημοσιογράφους. Δεν... Δεν είχα καμία απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Νάιτζελ Φαράζ οπότε ρωτήστε τον εκείνον εσείς απευθείας. Ε, Λίμπε Μπίργκιτ Σίπελ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση προ την Ελίζαμπεθ Ντένχαμ. Μπορείτε να μα εξηγήσετε και πάλι σε όλου του χρήστε ποια στοιχεία ακριβώ επεξεργάζεται το Facebook. Είναι αυτά του λογαριασμού, είναι με τα δεδομένα. Και αυτό που λέει aggregated gate data το Facebook αυτά δίνονται στις άλλες εταιρείες όπως η Cambridge Analytica και άλλες και καθώς μάθαμε από τις συσχετήσεις τα προφίλ και αυτά τα ομαδοποιημένα στοιχεία δεδομένα μπορούν εύκολα να ε, αναλυθούν για να χειραγωγήσουν κόσμο και να αγοράσουν ακόμα και ψήφου ε, χρησιμοποιώντας τα προφίλ, πράγμα το οποίο βλάπτει βασικού πυλώνε τη δημοκρατία μα. Πώ, ε, λοιπόν ε, το GDPR μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καθώ και το μελλοντική νομοθεσία περί ιδιωτικής ζωής, ιδιωτικότητα, θα χρησιμεύσουν. Αυτό είναι τμήμα της έρευνάς μας. Ακριβώς ποια δεδομένα πήγαν πού, από ποιον και ποια ήταν η ροή μέσα από ολόκληρο το σύστημα, πώς συνδυάστηκαν αυτά τα δεδομένα με άλλα δεδομένα από άλλους ε, ενδιάμεσους που χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Ε, τεράστιος είναι ο όγκος, εκατοντάδες τεραμπάιτ δεδομένων για να δούμε ακριβώς την ροή, την τροχιά των δεδομένων, αλλά θα φτάσουμε μέχρι το κόκκαλο και ε, θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα μέσα στην έκθεσή μας. Τώρα, όσον αφορά το GDPR, ήδη περιλαμβάνει αρκετές αρμοδιότητες ώστε οι αρχές προστασίας δεδομένων να μπορούν μπορούν να προχωρήσουν και να παρακολουθήσουν το μονοπάτι που ακολουθούν τα δεδομένα, να μπορούν να εξετάσουν in situ αλγόριθμους ενώ λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα για να δουν ακριβώς τι κάνουν επιτόπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ε, να κάνουμε ευνίδιους ελέγχους, να εξετάσουμε τους χώρους, τις υποδομές, να δούμε πώς στείνονται αυτές οι ροές δεδομένων και να τις παρακολουθήσουμε μέσα από όλο το σύστημα. Το GDPR είναι μια καλή αρχή και είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται. Κυρία Στίβενς από το ECR. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της σημερινής συνεδρίαση είναι το σκάνδαλο του Facebook και της Cambridge Analytica, αλλά δεν είμαι τόσο βεβαία αν θα πρέπει τεχνητά να περιοριστούμε σε αυτήν μόνο την υπόθεση. Εφόσον ε, ε, εγώ απευθύνομαι στην εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, την Επίτροπο για την πληροφόρηση. Πρόκειται για το μόνο σκάνδαλο ή υπάρχουν και άλλα μικρότερου διαστάσεων ε, σκάνδαλα. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν δεδομένα και τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια των ατόμων που, στους οποίους ανήκουν αυτά τα στοιχεία. Χωρίζεται τη συνένεση δηλαδή. Και ένα δεύτερο κομμάτι στην ερώτηση ερώτησή μου είναι πιστεύετε πως ο κανονισμός GDPR θα αλλάξει κάτι ή θα επιβληθεί στους μικρότερους παίχτες ενώ οι μεγάλοι θα μπορέσουν να το παρακάμψουν πιο εύκολα. Ξέρω πως ένας προηγούμενος συνάδελφος έστεσε αυτή την ερώτηση, αλλά θέλω συγκεκριμένη απάντηση γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Σας ευχαριστώ. Elizabeth Denham. Εσείς με ρωτήσατε αν πιστεύω πως αυτού του είδους η δραστηριότητα για την οποία μιλάμε σήμερα με το Facebook και την Cambridge Analytica συμβαίνει και σε άλλες πλατφόρμες αν δεν υπάρχουν άλλες εφαρμογές ή ε, ε, κατάχρηση και κακή χρήση προσωπικών δεδομένων. Λέω ναι, ε, και στον πολιτικό στίβο υπάρχουν και άλλες συμβουλευτικές εταιρείες που συνεργάζονται με συλλέκτες δεδομένων και εταιρείες ανάλυσης δεδομένων. Υπάρχει γενικά έλλειψη διαφάνειας για τους χρήστες σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Το Facebook όμως είναι πολύ μεγάλος φορέας εδώ, πολύ μεγάλος παίκτη και γι' αυτό και είναι η, έμφαση δίνεται σε αυτόν ε, στο Facebook για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, συμβαίνει και αλλού. Οι αρχές προστασία δεδομένων, οι βουλευτές, οι χρήστε, ε, οι υπερασπιστέ, οι δημοσιογράφοι ε, το γνωρίζουν τι συμβαίνει. πολύ σημαντική στιγμή για την προστασία δεδομένων. Η δεύτερη σα ερώτηση αφορούσε αν το GDPR θα αλλάξει κάτι ή αν θα βαρύνει μόνο τι μικρέ επιχειρήσει. Εγώ νομίζω πως ο γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων σημαντικό βήμα. Είναι ένα βήμα, αλλά θυμηθείτε, αυτή η νομοθεσία έχει γραφτεί στο χαρτί. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η επιβολή αυτής της νομοθεσίας στην πράξη. Δηλαδή είναι οι δραστηριότητες τις οποίες θέλουν, θα θελήσουν να κάνουν οι αρχές προστασία δεδομένων, είναι οι κυρώσει, τα πρόστιμα, οι χρήστες και οι πολίτες να καταλάβουν αρκετά καλά τα δικαιώματά τους για να προβούν σε δράση. δεν έχουμε χιλιάδες επιθεωρητές και υπόπτες που θα ελέγξουν ένα ένα τα συστήματα, ενώ έχουμε εκατομμύρια χρήστες, εκατομμύρια πολίτες που μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η επιβολή και η διαχείριση αυτής της νομοθεσίας θα είναι σημαντική. Θα πάρει κάποιος, ε, κάποιο καιρό για να εφαρμοστεί και το GDPR δεν είναι κατά των μικρών. Ε, νομίζω πως οι αρχές προστασία δεδομένων θα δράσουν ανάλογα, αναλογικά στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν την νομοθεσία και σίγουρα αυτό ισχύει για τη δική μας ε, εποπτική αρχή. Η Σόφη Ιντεβελτ τώρα από τους φιλελεύθερους, ε, από την Επιτροπή Λίμπη, Προς τον κύριο Γουάιλι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσλάβει μια εταιρεία για το project ε, της Ευρωπαϊκής ε, Διαλειτουργικότητας. Η εταιρεία αυτή ωστόσο έχει, ε, είναι συνεταίρος της CIA. Νομίζετε πως είναι, και έχει επίσης συνεργαστεί με την Cambridge Analytica. Και ο πρέσβης τον είπα στη Γερμανία δήλωσε χτες ότι θέλει να βοηθήσει τις συντηρητικές δυνάμεις να κερδίσουν τις εκλογές στην Ευρώπη. Τι θα κάνει η ΑΕΣΙΟ για να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν παράνομες μέθοδοι και θα δράσει αρκετά γρήγορα εάν και εφόσον παρέμβει. Δύο, σε δύο απευθύνατε την ερώτησή σας, ε, Σόφη. Ο κύριος Γουάλι... Ναι. Εσείς με ρωτήσατε για την εταιρεία Palantir που, είναι, που συνεργάζεται με τη Δυσία και με την Cambridge Analytica. Ναι, ε, υπήρξαν ε, ε, υπάλληλοι της Palantir που έχουν έρθει και έχουν εργαστεί σε πολλά από τα project που εγώ σας περιέγραψα όσο ήμουν εκεί. Μάλλον δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να σας πω, να πω στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με ποιον θα πρέπει να συμβληθούν, αλλά αυτό που σίγουρα θα σας πω είναι ότι Επειδή μια εταιρεία εργάζεται σε ένα θέμα και μια άλλη επισήμως εργάζεται σε κάποιο άλλο, δεν σημαίνει πως το προσωπικό τους προσωπικά δεν εργάζεται και για τα δεδομένα και δεν μοιράζεται πληροφορίες, δηλαδή υπό, υπόγεια, ας το πούμε. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί που θα εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε εταιρεία εργάζεται για ένα project θα είναι διαφανής για το με ποιους συνεργάζεται, αλλά και το τι κάνουν οι υπάλληλοι της ε, από δίπλα. Ε, καλές ερωτήσεις. Γι' αυτό ε, κατ' εξαίρεση να αφήνω δύο ε, προσώπους, δύο να απαντήσουν. δεν είναι η ευθύνη του ICO και όλων των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας των δεδομένων να επαγρυπνούν συνέχεια και μόνο, αλλά το θέμα είναι οι αλγόριθμοι και οι πηγές των δεδομένων και σύμφωνα με το GDPR και τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορέσουμε να ε, κάνουμε κοινοποιήσεις ε, επιβολής ε, ώστε να αναγκάσουμε τις εταιρείε να διαγράψουν αλγορίθμους ή να σταματήσουν να επεξεργάζονται δεδομένα. Και νομίζω ότι αυτές οι τα εντάλματα για την πάυση της επεξεργασίας θα είναι πιο ισχυρά από οποιαδήποτε διοικητικά πρόστιμα. Η κυρία Σπινέλη, ένα λεπτό. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Καρόλ Κατβαλάντρο. Να πάω αντίθετα με το ρεύμα. Αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα της Cambridge Analytica και των λοιπόν ο Κρίστοφερ Βάιλι υποστηρίζει ότι η στόχευση των χρηστών βασιζόταν στους εστερικούς τους δαίμονες και έτσι επηρεάστηκε η Αμερικανική ψηφοφορία και το Brexit. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες αλλά αξιόπιστες αναλύσεις λένε ότι η επίδραση ήταν ελάχιστη. Πολύ μικρότερη από αυτήν που λέγεται. Λένε ότι το μικρό targeting έγινε χωρίς συνένεση από τον Ομπάμα το 2008 και το 2012 και ότι ενθουσίασε τις ε, κύριες εφημερίδες. Ο χρήστης καταναλωτής συγχέεται με τον ε, ψηφοφόρο. Ωστόσο, οι δύο αυτοί έχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Η Cambridge Analytica υποστηρίζει, ε, υποστήριξε τον Ted Cruz, αλλά απέτυχε. Αναρωτιέμαι κατά πόσο οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το σκάνδαλο αυτό για να αποφύγουν την ανάλυση των δικών τους ητών. Ευχαριστώ. Carol, please. Oh, for έχετε δύο λεπτά. Εκτός μικροφώνου μιλήτρια. Πολύ καλή ερώτησή σας για το πόσο αποτελεσματικές ήταν τεχνικές αυτές και είναι. Το ευρύτερο ερώτημα είναι όμως αν ήταν νόμιμες. Αυτό που επαναλαμβάνω διαρκώ όταν έρχεται ο κόσμο και μου λέει ότι όλοι το κάνουν αυτό, όλε οι πολιτικέ εκστρατείε, όλε οι προεκλογικέ εκστρατείε. Δεν ξέρω αν άλλε προεκλογικέ εκστρατείε που χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε, χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε ενό αναδόχου στρατιωτικού. Η ΕΣΕΛ έχει εργαστεί για τη Βρετανική κυβέρνηση, για το Υπουργείο Άμυνα. Έχει αμυφθεί από τη Βρετανική κυβέρνηση για ασκήσεις προπαγάνδας σε χώρε. αλλού. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι έχουν κάνει γιατί ήταν απόρριτο. Οι τεχνολογίε του, οι τεχνικέ που χρησιμοποιούν ε, εξελίχθηκαν μέσω αυτών των δραστηριοτήτων και μετά στράφηκαν κατά του εγχώριου πληθυσμού. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Μπορεί να το συζητήσει ο κόσμος, αλλά δεν εστιάζομαι εγώ εκεί. Εγώ εστιάζομαι στο κατά πόσο έγινε αυτό νόμιμα, αν ήταν νόμιμο, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, ποιο τα δαπάνησε, σε τι και γιατί υπήρξαν οι συνδέσει όλες μεταξύ όλων αυτών των εταιριών και όλων αυτών των εκστρατιών και γιατί αποκρύφθηκαν. Για ποιο λόγο έμειναν κρυφέ οι σχέσει αυτέ. Και αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί υπάρχει και κάποιο άλλο εδώ που θα μπορούσε να σα δώσει κάποιε απαντήσει. Έχετε εδώ τον του UKIP, το UKIP έδωσε δεδομένα στην Cambridge Analytica που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος και το UKIP από ό,τι κατάλαβα ε, δεν ε, συμμορφώνεται με όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε εμεί ερωτήσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εσείς μπορείτε όμως, μπορείτε λοιπόν να τους ρωτήσετε, να τους κάνετε τέτοιες ερωτήσεις σε βάθος να μας εξηγήσουν. Ευχαριστούμε. Okay. Okay. Um, Libe ε, Λίμπε για του πράσινου είναι ο κ. Γιάνν Άλμπρεχτ. Παρακαλώ. Λοιπόν, να προσπαθήσω τώρα και εγώ να μεταφέρω τι ερωτήσει αυτέ προς ε, τον κύριο Βάιλι, γιατί ακριβώ πρέπει να δούμε τα γεγονότα τη υπόθεση. και θα ήθελα να καταλάβω ποιο ήταν ακριβώς το μοντέλο της Cambridge Analytica παραδείγματο χάρη στο δημοψήφισμα του Brexit με βάση ποια μοντέλα δεδομένων και επίσης ε, έχουμε και την ε, θυγατρική της την Aggregate IQ και την εμπλοκή της σε αυτές τις εκστρατείες ποια είναι τα μοντέλα δεδομένων, με ποια δεδομένα εργαστήκατε και ποιο ήταν το μοντέλο της ε, στόχευσης, γιατί αυτό πρέπει να αντιληφθούμε λίγο το πώς ε, συνέβη η διαδικασία. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Λοιπόν, ε, είναι δύσκολο βεβαίως να μπω σε λεπτομέρειες λόγω του χρόνου. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μπορείτε να δείτε τα πολλά στοιχεία της βιβλιογραφίας που βασίζονται στην εργασία της Cambridge Analytica. Οι εργασίες αυτές, κάποιες από αυτές, χρηματοδοτήθηκαν από την DARPA, το ερευνητικό κομμάτι του Αμερικανικού Πενταγώνου. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του ε, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον ε, είδα παραδείγματο χάρη κάποια ελεγχόμενα πειράματα που έδειξαν κάποια αλλαγή η πυθόε εάν θέλετε όσον αφορά τις συγκρίσεις με την ε, εκστρατεία του Ομπάμα χρησιμοποιήθηκαν πράγματι δεδομένα αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο για την χειραγώγηση των ψηφοφόρων και δεν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την παραπληροφόρηση. Οπότε Ναι, Δυστυχώ δεν μου επιτρέπει και ο χρόνος να επέκταθω στο πώ δουλεύουν τα μοντέλα, γιατί χρειάζεται περισσότερη ώρα. Ζητώ συγγνώμη, ε. έχουμε αυτού τους περιορισμούς. Ε, μπορείτε να επεκταθείτε με κάποιον άλλο τρόπο. Για την Λίμπε λοιπόν και την ΑΦΚΟ και το FTD ο Μπάτον. Ευχαριστώ Κλοντ. Εγώ τα τελευταία 26 χρόνια είμαι στην πολιτική και προσπαθώ να πείσω τον κόσμο ότι έπρεπε να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήμουν ε, κατά τέτοια της εκστρατείας και συνάντησα χιλιάδες ανθρώπους ε, πρόσωπο με πρόσωπο. Και κανένας ε, τότε, ούτε έκτοτε, μου είπε ότι με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάστηκαν από το οτιδήποτε είδαν στα κοινωνικά μέσα. Η υπόθεση αυτή είναι το ότι το κατεστημένο κάνει ό,τι μπορεί για να αναστρέψει την απόφαση του δημοψηφίσματος. Και η ερώτησή μου είναι προς την κυρία του Guardian, ο οποίος βεβαίω δεν είναι αμερόληπτος, αλλά έχει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, όπως και οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή ε, καμπάνια. Η καμπανια η ερωτηση μου είναι, ο Guardian έχει ερευνήσει την εκστρατεία που έλεγε να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο με τον ίδιο τρόπο που ερευνά την εκστρατεία για να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεύτερον, η στάση των Guardian μήπως είναι τελείως κομματική για να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί να αναστραφεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. δεν είναι το θέμα παρταξιακό. Το θέμα αφορά την ακαιρεότητα της δημοκρατίας μας, αφορά την εθνική κυριαρχία και νομίζω ότι ε, και εσάς ε, θα σας ενδιαφέρε κάτι τέτοιο. Για να έρθω στην ερώτησή σας. Εάν ο Guardian ερευνά την χρήση δεδομένων ε, της άλλης πλευράς. Δεν γνωρίζω τέτοια ζητήματα από την άλλη πλευρά. Δεν ε, έχω συναντήσει κάτι και δεν νομίζω ότι και η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει συναντήσει κάτι τέτοιο ή να ερευνάει η αστυνομία κάτι. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ελπίζω ότι θα το αποκαλύψουν οι δημοσιογράφοι και θα ερευνηθεί. σημαντικό να έχει νομίζω σημασία το ποιος διαπράττει τα εγκλήματα ή προσπαθεί να ανατρέψει την εκλογική νομοθεσία, αλλά να λογοδοτεί στην δικαιοσύνη. Και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε πλήρω. Το για το ότι πρόκειται για κάτι το παραταξιακό η, η έρευνα την οποία κάνουμε. Δεν νομίζω ότι το Facebook ή η Google έχουν κάποια πολιτική ή παραταξιακή τοποθέτηση επηρεάζουν χώρες και δημοκρατίες όλων, όλου του πολιτικού φάσματος ανά τον κόσμο, σίγουρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι εάν θέλετε να θάβετε το κεφάλι σας στην άμμο και να θεωρείτε ότι είναι το κατεστημένο του Remain, εντάξει, τι να πω. Συνεχίστε έτσι. Πραγματικά πρέπει λίγο να σκεφτείτε παραπέρα και να δείτε την ευρύτερη εικόνα και τον ευρύτερο κίνδυνο. για την ΙΜΚΟ και το ΙΕΝΕΦ ε, ο κύριος, ε, η κυρία Μελίν Τρουσίνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σαν αυτή του κύριου Μπατέν, οπότε θα επικεντρωθώ σε ένα τεχνικό ερώτημα. Κανονικά θα μπορεί να την απαντήσει ο κύριος Παρακύλας. Ε, εσείς το αποφασίσετε. Λοιπόν, εγώ αντιλήφθηκα ότι έχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση της προστασίας δεδομένων το Facebook μετά από μια επίσκεψη που έγινε πριν στο φθινόπωρο. Η συλλογή πληροφοριών από τις πλατφόρμες ε, ε, κοινωνικών ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται βάσει αλγορίθμων με τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προεκλογικές εκστρατείες αλλά όχι μόνο. Η εμπορική χρήση των προσωπικών μας δεδομένων είναι ανατριχιαστική ενίοτε. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μερικές φορές στο facebook οι άλλοι μας ακούνε ή διαβάζουν τα email μας. Έχω λοιπόν μια τεχνική ερώτηση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των τεχνικών εκμετάλλευσης που χρησιμοποιήθηκαν ε, κατά την εκστρατεία του Τραμπ ή του Brexit και εκείνων που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους. Σάντι. Πιστεύω ότι η βασική ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχει διαφορά μεταξύ των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην προεκλογική στρατεία του Τραμπ και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Η απάντηση είναι όχι. Στην εκστρατεία του Τραμπ χρησιμοποιήθηκαν πολύ αποτελεσματικά οι εμπορικές ε, τεχνικές και οι τεχνικές μάρκετινγκ που έχουν αναπτυχθεί για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια για τους σκοπούς μιας πολιτικής εκστρατείας και μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν πολύ αποτελεσματικά. Ήταν ε, ίσως ε, η πιο αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία που έχουμε δει ποτέ για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστούμε για τη ΛΥΜΠΕ και το ΕΛΚ. Κύριε Νάγκε, έχω μια σύντομη ερώτηση. Η κυρία Γιαρόκα, ήθελα να επανέλθουμε στο κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε τι οικονομικό κέρδος αποκόμισε το Facebook, υπήρχαν τρίτα μέρη. Ήθελα επίσης να μάθω, συμβαίνουν αυτά και σε άλλες χώρες, πολιτικές εκστρατείες, ε, έτσι, οι κυβερνήσεις ε, που πληρώνουν για να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνικές. Αν χρησιμοποιείτε λέει δηλαδή, τέτοιες τεχνικές σε πολιτικές εκστρατείες ή σε ε, κυβερνήσεις σε άλλες χώρες. Ποιος θέλετε να απαντήσει. Εκτός μικροφώνου ομιλήτρια. Θα δούμε η κυρία ε, Κάλε Βόλτερ δεν θέλει να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ να απαντήσω εγώ. Τον κύριο Ντέβιτ τον έχουμε αφήσει λίγο απ' έξω, παρακαλώ, μην τον ξεχνάμε. Τον κύριο Ντέβιτ Κάρολ. Λοιπόν, ρωτήσατε τα κέρδη των πολιτικών εκστρατιών και κατά πόσο εμπλέκονται τρίτα μέρη και ποιο είναι το κέρδος του Facebook. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο γενικά εδώ, διότι το Facebook δεν ανακοινώνει δημοσίως τα οικονομικά του για πολιτικές εκστρατείες γενικότερα ή ούτε για ειδικότερε ε, άλλες εκστρατείες. Δεδομένων αυτών, ενίοτε εμπλέκονται τρίτα μέρη στην ε, εφαρμογή μιας ε, εκστρατείας marketing στο Facebook και αυτά τα μέρη λαμβάνουν κάποιο κομμάτι του ποσού. Αλλά γενικά η πλειοψηφία η, όλων των χρημάτων που δαπανώνται από το Facebook, ε, στο, συγγνώμη, στο Facebook για διαφημίσεις πάει στο Facebook. Ο αριθμός που έχουμε για την εκστρατεία του Τραμπ για, την για τις προεδρικές εκλογές ήταν ε, της τάξης των 80-90 εκατομμυρίων ε, δολαρίων Αμερικής, για να καταλάβετε τη κλίμακα. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους αν φύγετε και έχει έρθει η ώρα σας για να κάνετε ερώτηση, έφυγε, δεν έχετε μετά τη δυνατότητα. Κυρία Καϊλή, για τους σοσιαλιστές, η κυρία Καϊλή, Ήθελα να στραφώ στο... να ρωτήσω για το Facebook. Είναι δυνατό να διαγράψουμε τα δεδομένα μας, να τα εξάγουμε, να τα δούμε ποιος χρησιμοποίησε τι, ποιος ε, έδωσε πρόσβαση σε τρίτα μέρη, σε ποιους, κατασκευαστέ συσκευών. Ουσιαστικά μπορούμε να μην δίνουμε τα δεδομένα μας όλα αυτά, αλλά να μπορούμε να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές. Έχετε μετρήσει επίσης ε, πώς ε, ε, ε, επηρεάζεται το περιεχόμενο, οι ειδήσει με κάποιο τρόπο ή όχι. Τέλος πιστεύετε ότι τα συνολικά δεδομένα, η συγκέντρωση δεδομένων πρέπει να αποτελέσουν δημόσιο αγαθό για την επιστήμη. Έχετε ιδέες, έχετε προτάσεις ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Επειδή η νομοθεσία όπως το GDPR καθυστερεί λίγο, δεν δίνει τη δυνατότητα ε, στο να γίνει, ε, να υπάρχει καινοτομία για τη στοχευμένη ε, διαφήμιση χρειάζονται κανόνας. Επειδή αναφέρετε το Facebook, να σου πω ότι δεν δουλεύουν πια για το Facebook, δεν δουλεύουν για αυτές τις εταιρείε εδώ. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Πολλά είπατε. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω. Η πρώτη πτυχή είναι ο έλεγχος που έχουν οι χρήστες. Λοιπόν, το Facebook, λόγω του ότι υπόκειται σε διάφορε νομοθεσίες και στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, έχει διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, ένα από τα πράγματα που προέκυψε επανελειμμένος είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι έλεγχοι αυτοί δεν λειτουργήσαν όπως ε, είχαν σχεδιαστεί να λειτουργήσουν. Μια συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί είναι αυτό που αναφέρατε εσείς ε, για τους κατασκευαστές ε, κινητών συσκευών που έδωσαν ιδιωτική πρόσβαση σε δεδομένα. Η ρύθμιση που δεν λειτουργήσε ήταν μια ρύθμιση που έχουν οι χρήστες για να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση στα δεδομένα τους από φίλους. Οι New York Times έκαναν έναν έλεγχο λοιπόν αυτής της ρύθμισης να, για απενεργοποίηση της πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα δεδομένα διαβιβάστηκαν ούτως ή άλλως. Εδώ έχετε ένα παράδειγμα ρύθμισης που δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. ένα από τα βασικότερα θέματα του διαταγμάτου της στις ΗΠΑ. Το δεύτερο αφορά τη ροή ειδήσεων και πώς ε, επιλέγετε συγκεκριμένο περιεχόμενο και τι μας απασχολεί εκεί. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε για τη ροή ειδήσεων είναι ότι προσπαθούν να επιλέξουν ταυτόχρονα το καλύτερο ε, περιεχόμενο που θα θεωρήσουν οι χρήστες ενδιαφέρον αλλά και το οποίο ταυτόχρονα θα βοηθήσει το Facebook και τι άλλες να βγάλουν χρήματα. Έχουν λοιπόν σχεδιάσει τι ροέ ειδήσεων ώστε να είναι ελκυστικέ. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει πολλή χρόνο, θα απαντήσω πολύ γρήγορα το ε, σύνολο δεδομένων, τα σύνολα δεδομένων που αναφέρατε. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα δεδομένα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο να το απαντήσω πέντε δευτερόλεπτα. Αλλά σίγουρα τα συγκεντρωμένα δεδομένα, ε, ανάλογα με το πόσο εύκολα μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα, είναι κάτι το οποίο θα ε, έχουμε να εξετάσουμε στο μέλλον με πολλέ προσπάθειε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για εμένα το βασικό ερώτημα είναι πώς θα μετακινηθεί η ισχύ από τις πλατφόρμες ε, ξανά στους ανθρώπους για να έχουμε εκπροσώπους που τη δίκαια και δίκαια αποτελέσματα δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα μου λοιπόν απευθύνω στον κύριο Παρακύλας. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ λέει πως αντιμετώπισε τις αδυναμίες, όμως γνωρίζουμε ότι τα βασικά στοιχεία οι αλγόριθμοι, οι στοχευμένες διαφημίσεις, η τεχνολογία πίθους ε, εξακολουθούν να παραμένουν. Οπότε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κατάχρηση την επόμενη φορά και τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε αποτελέσματα όπως το Brexit που εμένα μοιάζει η ληστεία του αιώνα. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν λοιπόν διαφορές πτυχές που πρέπει να δούμε και από την πλευρά των εταιριών και από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Από την πλευρά των εταιριών νομίζω ότι το Facebook κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα τώρα ε, και εφαρμόζει την διαφάνεια στην διαφήμιση για να καταλάβουμε ποιος αγοράζει ε, διαφημίσεις ε, για τις εκλογές. Ένα σημαντικό βήμα, αν και βεβαίως δεν είναι όλα όσα πρέπει να γίνουν ακόμα για να υπάρχει διαφάνεια. Όμως ένα σημαντικό πρόβλημα στην πλευρά αυτών των εταιριών είναι ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι να συλλέγουν όσο δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να προσφέρουν πολύ στοχευμένες διαφημίσεις και να πουλάνε μετά αυτές τις διαφημίσεις ε, στον πλειοδότη και έτσι δημιουργούνται κάποια κίνητρα επικίνδυνα. Αυτή είναι η απλή αλήθεια όσον αφορά αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Υπάρχουν λοιπόν δύο προσεγγίσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε εδώ. Είτε να ρυθμίσουμε όλες τις χειρότερες ε, περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη ξένες δυνάμεις που θα ευλέκονται σε εκλογές και να λέμε τι πρέπει να γίνει με πολύ πολύπλοκους κανόνες ή να αφαιρέσουμε κάποιες από τις λειτουργίες για να υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες στόχευσης, για να είναι δυσκολότερο να γίνουν αυτά τα οποία συνέβησαν στο Brexit και στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Αυτές είναι οι δύο βασικές ε, προσεγγίσεις. Εγώ θα σας ενεφάρει να αποφύγετε πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Ε, δηλαδή δεν μπορείτε να γράφετε πράγματα όπως ε, οικοσυστήματα και κίνητρα και προσπαθήστε να βρείτε και άλλους παίκτες στα οικοσυστήματα που θα μπορούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι πολύ συγκεκριμένη η απάντηση, αλλά είναι περίπλοκο το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τρίτη φορά, με τρίτη ιδιότητα, η κυρία Σπινέλη για την κουεπίτε μας λοιπόν, γιατί ακριβώς μιλάτε. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Σάντι, τον παρακυλασσά στα Ιταλικά. Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους πολίτες. Τι ρωτάω, αυτός ο πολλαπλασιασμός των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία μας ε, μπορεί να επηρεάσει ε, τις ελευθερίες και την πολυφωνία στο διαδίκτυο αρνητικά. Μπορεί επίσης να δυσκολέψει την πρόσβαση. Δηλαδή έχουμε τον πόλεμο στα fake news, τους νόμους προστασίας του copyright, προστασίας ε, νόμους διοντολογίας, κώδικες διοντολογίας για την αφαίρεση κάποιων περιεχομένων. Η εντύπωσή μου είναι ότι προσπαθούμε να ξαναβάλουμε την οδοντόκρεμα μέσα στο σωληνάριο. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Συμφωνώ. Πράγματι υπάρχει μια οδοντόκρεμα και ένα πρόβλημα οδοντολογικό. Είναι δύσκολο να πάμε πίσω και να διορθώσουμε προϊόντα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει όταν κανείς δεν ήξερε ε, ποιες θα ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις όταν αγόρασε το προϊόν. Θα ενθάρρυνα λοιπόν και εσά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα να σκεφτείτε ευρέως το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κίνητρα για κάποιες εταιρείες ώστε να δρουν σωστά και να μην δρουν παράνομα. Αναφέρατε το GDPR, τον κανονισμό ένα από τα βασικά του στοιχεία είναι ότι περιλαμβάνει ε, σημαντικές ποινές κυρώσεις. Για πρώτη φορά οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται ενώπιον ε, πιθανότητας ε, σημαντικών οδυνηρών κυρώσεων και ποινών. Όταν αλλάζει κανείς την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας μέσω της απειλής ενός σημαντικού προστίμου, αλλάζει τις προτεραιότητες της εταιρείας ώστε να αποφύγει αυτή την κατάσταση με την οδοντόκρεμα που μόλις αναφέρατε γιατί δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά ε, ενώπιον ε, ενός προστήμου πολλών δισεκατομμύριων δολαρίων. Οπότε ξανασκεφτείτε τα οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα. Μην φοβάστε τις ποινές, μην φοβάστε τα πρόστιμα, αλλά έχετε στο νου σας και τις μικρές εταιρείε ώστε να τις προστατεύετε. Τις μικρές εταιρείε που κάνουν καινοτόμα πράγματα, καλά πράγματα, χωρίς να τους ρίχνουμε την ευθύνη των μεγάλων εταιριών που δημιουργούν ξαφνικά αυτές τις ε, κοιλίδες που αναφέραμε. Ευχαριστούμε για τους πράσινους, η Τζούτιθ Αργεντίνη. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Καντ Βαλάντερ. Ήθελα να μιλήσω για την επιρροή του Κρεμλίνου στο δημοψήφισμα του Κρεμλίνου. Εγώ είμαι από την Ολλανδία, είχαμε και εμείς ένα δημοψήφισμα για την Ουκρανία και για μας τέθηκε το θέμα της ε, επίδρασης ε, ε, των εκστρατιών κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματο εκείνου στις κατοχώρες και μα ανισχύει. Μας ανισχύει όλους. Ήθελα να, να καταλάβω πόσο πιστεύετε σημαντική ήταν η επίδραση τη Ρωσία στην εκστρατεία ε, αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι κύριοι παράγοντε. Από ό,τι κατάλαβα επίση, εσείς ε, λάβατε προσωπική επίθεση εκεί. Είστε ασφαλείς εσεί προσωπικά. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι το βασικό εδώ ε, είναι ότι δεν ξέρουμε. Η υποψία βεβαίως είναι ότι η Ρωσία επηρέασε με κάποιον τρόπο το δημοψήφισμα του Brexit. Γιατί γνωρίζουμε ότι ε, επηρεάζει τις εκλογές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φαίνεται πως ε, σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία θα ήταν απίθανο να μην προσπαθούσε. Αλλά και πάλι βεβαίως το θέμα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και αυτό το οποίο είπα πριν. Αυτό το οποίο δηλαδή μοιάζει με συστημική ε, αδυναμία του να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το οποίο όντως γνωρίζουμε είναι ότι το Facebook εμποδίζει τις σχετικές προσπάθειες ε, στα αιτήματα δηλαδή του Ντέμιν Κόλλινς επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Το Facebook ε, έγραψε μια επιστολή τα Χριστούγεννα και είπε ότι κοίταξαν τους γνωστούς λογαριασμούς ε, από την υπηρεσία έρευνα του ίντερνετ και είπαν ότι ξοδευτήκε ένα δολάριο κατά τη διάρκεια του δημοψήφισματος και μετά πριν από τρεις εβδομάδες ε, το Κογκρέσο δημοσίευσε όλες αυτές τις διαφημίσεις είδαμε αυτές που στόχευαν και την Βρετανία και εκεί πέρα είδαμε ότι υπήρχαν πάνω από χίλιες λίρες που είχαν εξοδευτεί και πάλι εντάξει δεν ακούγεται μεγάλο ποσό, αλλά είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα δολάριο. Αυτή ήταν λοιπόν η πολύ στενή ερμηνεία του Facebook. Αλλά... Λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερα και πρέπει να μας βοηθήσετε γιατί η Βρετανία παλεύει με αυτά τα ερωτήματα και χρειαζόμαστε την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ για την ΑΦΚΟ και το ευθύτιο κύριο Ζουλού. Χαίρετε. Ερώτησή μου απευθύνεται στον Σάντι Παρακύλα. Σήμερα μιλήσαμε για το GDPR που είναι σίγουρα ένα βήμα μπροστά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη συζήτηση προέκυψαν διάφορες λύσεις για να προοδεύσουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την νομοθεσία, δηλαδή να ζητήσουμε τη διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων, να βλέπουμε καλά τα περάσματα από τον ένα φορέα στον άλλο... να ζητήσουμε περισσότερες εξουσίες για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε αποδεικτικά στοιχεία και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Σήμερα στην ΙΜΚΟ ψηφίσαμε και για την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων και εδώ θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή γιατί όταν μιλάμε για μη προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα ένα μήνυμα που στέλνουμε δεν είναι προσωπικό δεδομένο αλλά λέει πολλά για μας. Υπό το φως της εμπειρία σας, ποιο άλλη πρόταση θα μπορούσατε να μας δώσετε για την ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη των υγιών εταιριών και έπειτα αυτά τα νομοθετικά πλαίσια κυρίως ε, να μπορούν να, να, μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες επιχειρήσεις και να μην επιβαρύνουν τις μικρές. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω πως ε, τα κεντρικά θέματα που, επαναλαμβάνω, που θα επαναλάβω είναι τα, αυτά που είπα και στην αρχική μου ομιλία. Δηλαδή να σκεφτούμε κίνητρα, να σκεφτούμε την προστασία των μικρότερων εταιριών, και νομίζω πως αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Μπορείς να τις εξαιρέσεις από ορισμένου κανόνες, ας πούμε, ανάλογα με τους κανόνες. Μπορείς να περιορίσεις τις ποινές. Μπορείς επίσης να σκεφτείς την ε, εκπαίδευση και την υποστήριξη. Ίσως αυτό είναι ένας τομέας που δεν είναι απαραίτητα πρώτη σκέψη του καθενό, Πάντω, αν κανείς θέλει να συμμορφωθεί με το GDPR και το είδαμε πολύ κόσμο που γνωρίζω στο GDPR, που, που ξοδεύουν πολύ, κόσμο, ε, πολύ χρόνο και προσπάθεια για να συμμορφωθούν στο GDPR, Μπορεί να υπάρξει λοιπόν στήριξη όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και πόροι ώστε να βοηθηθούν οι μικρές εταιρείες. Τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτές λοιπόν να συμμορφωθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι πέρα από τα όσα ήδη είπα τα βήματα, ίσως αυτός και να, να είναι ένας τομέας όπου εγώ θα επεκτηνόμουν περισσότερο. Δηλαδή να σκεφτείς καλύτερα για το πώς μπορείς να βοηθήσεις τις μικρές εταιρείες πέρα από την μείωση των ποινών. Πώς μπορείς πρακτικά να τις βοηθήσεις πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσουν να συμμορφωθούν ε, βοηθούμενες και από πόρους που μπορείτε να προσφέρετε. Άξελ Φως, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παρακυλές. Αν δείτε την περίπτωση αυτή, εντάξει, στην αρχή σοκαριστήκαμε και μετά ο συνήθως λέμε χρειάζονται αυστηρότεροι νόμοι κτλ. κτλ. Θα ήθελα να μου πείτε, ακούγοντας ε, τις απαντήσεις ε, και της κυρίας Σεντεναμ και του κυρίου Τζόνστον, ότι τελικά απαιτείται περισσότερος έλεγχος και εφαρμογή αντί για περαιτέρω νόμοι και κανόνες ή έχουμε ξεπεράσει αυτό το σημείο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει ακόμα κατά την αποψή σας τεχνικά, νομικά ή πολιτικά για να αποφευχθούν τέτοιες καταχρήσεις ε, ανθρώπων ή εκλογών για να εμποδιστούν αυτά τα φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε για την πρώτη ερώτηση για την επιβολή των υφιστάμενων νόμων. Ε, δεν είμαι ειδικό εγώ στην Ευρωπαϊκή Προστασία Δεδομένων, αλλά οπωσδήποτε στις ΗΠΑ δεν εφαρμόζεται ούτε η υφιστάμενη νομοθεσία. Ε, Παραδείγματο χάρη η νομοθεσία περί συνένεσης. Δηλαδή, οπωσδήποτε το να διασφαλίζουμε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τους απαραίτητους πόρους και ενθαρρύνονται ε, ε, επιβάλλουν τον νόμο, νομίζω είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις νομοθεσία στην περίπτωση της ε, Cambridge Analytica. Όσον αφορά τους νέους κανόνες, νομίζω ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δομένων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα και θα πρέπει να γίνει σκέψη για την επόμενη γενιά της τεχνολογίας. Δηλαδή, ενώ ο γενικός κανονισμός κάνει μια πολύ καλή δουλειά για να αντιμετωπίσει κάποια από τα ζητήματα με τις ε, τρέχουσες τεχνολογίες. Το τι έρχεται είναι πραγματικά τρομοκρατικό. Δηλαδή η δυνατότητα να δημιουργηθεί περιεχόμενο το οποίο είναι πραγματικά τελείως ψευδές, ε, άνθρωποι που μοιάζουν να μιλάνε αλλά δεν έχουν πει ποτέ αυτά τα πράγματα. Ε, τεχνητή νοημοσύνη που προβλέπουν τις δράσεις των χρηστών πριν γίνει καν. Το Facebook είναι μία από τις εταιρείε που εργάζεται πάνω σε κάτι τέτοιο και σκεφτούνται πώς θα πωλήσουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τις μελλοντικέ δράσεις. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά το πλαίσιο αυτών των νέων τεχνολογιών. Και θα σας ε, ενεθάρει να τα δείτε πολύ γρήγορα αυτά τα ζητήματα. Για την ΛΥΠΕ και του Σοσιαλδημοκράτε ο κύριος Βάινχολτσερ. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Κατβαλάνδρο. Ευχαριστούμε για την ιστορία που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστούμε για την ε, αντοχή σας, την επιμονή σας. Ε, αγγίζετε τις καρδιές, ε, την καρδιά των δημοκρατικών κοινωνιών μας. Πώς θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους από ξένη επίδραση. Το είδαμε στο πλαίσιο του Brexit, πώς επηρεάστηκε το μέλλον. Και η ερώτησή μου είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε την επιβίωση των δημοκρατιών μας. Για να το πω τόσο απλά προστατεύοντας ε, τους πολίτες από οποιοδήποτε είδους εκλογική χειραγώγηση. Και πού θεωρείτε ότι λείπει νομοθεσία ε, η έλλειψη επιβολής ε, υπαρχόντων κανόνων και εφαρμογής τους. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω και που θεωρειτε οτι λειπει νομοθεσια η ελλειψη επιβολης των κανονων και εφαρμογης τους ευχαριστω από την ερώτηση του κυρίου Μπάτον είπε ότι κανείς από όλους, όλους εκείνους με τους οποίους συζήτησε δεν θεωρεί ότι επηρεάστηκε από κάτι που διάβασε online και σίγουρα το θέμα στο δημοψήφισμα ήταν ότι πολλοί κόσμοι είχε μετακίνητες απόψει, αλλά πολύ λίγοι, ένα μικρό κομμάτι δεν είχε μετακίνητες απόψεις και το θέμα ήταν να βρεθούν αυτοί, αυτοί οι λίγες χιλιάδες άνθρωποι ουσιαστικά τους βρήκαν, τους εντόπισαν και τους βομβάρδισαν με πληροφορίες αυτό ήταν αόρατο σε όλους μας αυτό είναι που δεν είδαμε. Και αυτό είναι που συμβαίνει και σε εκλογές και στις δικές σας χώρες είμαι βέβαιη. Έχουμε λοιπόν ένα κόσμο καθησυχασμένο, ο οποίος θεωρεί ότι εμένα δεν με επηρεάζει αυτό, εγώ δεν το είδα, δεν με πειράζει εμένα, αλλά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα συμβαίνει ε, στα κρυφά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όλα αυτά έχουν συμβεί στα κρυφά. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό αυτό που κάνετε, ότι ε, φωτίζετε αυτές τις πρακτικές και βλέπετε ε, τι μπορείτε να κάνετε εσείς ώστε να διασφαλίσετε το μέλλον, μαθαίνοντας για παράδειγμα από όσα έμαθε α πούμε η Ελίζα από τις ερευνές της, διότι θεωρώ ότι το να εφησυχαζόμαστε όπως ακούμε από κάποια σχόλια εδώ, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Συγγνώμη, ε, κοιτώ τριγύρω και βλέπω όλο τον κόσμο με τα ακουστικά. Έχουμε τόσες πολλές γλώσσες εδώ, τόσες ε, πολλές ε, ε, διαφορετικές νοοτροπίες, χώρες. Ξέρετε, αυτές οι διαφημίσεις δεν είναι απλά πολιτικές πυροδοτούν μίσος, πυροδοτούν διάφορα πολιτικά μηνύματα. Είναι πολύ ευρύτερο. Και εδώ θα σοπάσω. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Θα ήθελα να είμαι ουδέτερος, αλλά ξέρετε, μου άρεσε πολύ η απάντησή σας. Λοιπόν... Επόμενος ε, για την ε, ε, την Επιτροπή Λίμπε και το ECR είναι ο κύριος Βόρκεν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων του Facebook. Βλέπουμε ότι σβήνονται διάφορες σελίδες και οι κανόνες με τους οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου διαφανείς. Υπάρχει τέτοια πρακτική, υπάρχουν κάποιοι σαφοί κανόνες ε, σχετικά με το τι κατεβαίνει και σβήνεται για να μην υπάρχει λογοκρισία στο facebook και αν έχετε ε, λίγο χρόνο μια ερώτηση προς την κυρία Ντέναμ. Ε, σε ποια άλλη εκλογική εκστρατεία είχαμε ανάλογες τέτοιες καταχρήσεις προσωπικών δεδομένων Ελίζαμπεθ, η πρώτη σας ερώτηση αφορούσε την, την παράνομη διαγραφή δεδομένων από το Facebook και πρέπει να μου δώσετε το πλαίσιο αν ήταν ε, οι πληροφορίες προφίλ κάποιου ή αν ήταν ε, αποδεικτικά στοιχεία ή διοικητικές πληροφορίες. Αλλιώς δεν μπορώ να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στη Mercedes Bresso. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την Κάρολη είναι η ερώτησή μου. Το πρόβλημα είναι ότι το Facebook είναι ε, ε, μια πλατφόρμα όπου συμμετέχει το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι ο πιο μεγάλος δημόσιος χώρος του κόσμου. Για όλους μας οι κανόνες ε, λοιπόν που διέπουν αυτή την πλατφόρμα είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον μας. Άρα λοιπόν ε, η δημοκρατία βασίζεται στην εκπροσώπηση, αλλά ο καθένας έχει τη δυσκολία πώς να βρίσκεται σε αυτόν τον παγκόσμιο χώρο. Ε, εγώ θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν πιστεύετε από τη μια πλευρά ότι αυτές οι πρόσφατες απόπειρες από το Facebook για αυτοπεριορισμό των καταχρήσεων των οποίων να έχουμε πέσει θύματα είναι σοβαρέ, αν και αν είναι επαρκή Από την άλλη πλευρά, επειδή πολλοί έθεσαν αυτό το ερώτημα, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν επιρροές και για άλλες εκλογές, ας πούμε πρόσφατες Ιταλικές εκλογές και πολλών άλλων χωρών και ένα δίκτυο ε, δημοσιογράφων ερεύνης διεθνές δεν θα μπορούσε αποτελεσματικά να ελέγξει και να αναχαιτήσει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Σας ευχαριστώ για αυτή σας την ερώτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Είναι ένας δημόσιος χώρος που χρησιμοποιείται από, τεράστι, από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλά αυτό είναι το θέμα κλειδί. Δεν είναι δημόσιος χώρος. Είναι ιδιωτικό κεντρικός χώρος μιας εταιρείας, ενός ομίλου. Και αυτό καθίσταται σαφές για οποιονδήποτε έχει πέσει θύμα κατάχρησης σε αυτές τις πλατφόρμες και νωρίτερα έτεθη ερώτηση για απειλέ που είχα δεχθεί και μπορώ να το χρησιμοποιήσω διότι έγινε, μου, έγινε μια απειλή από το live.eu δηλαδή την εκστρατεία του Nigel Farage εναντίον μου στο Twitter όπου απειλήθηκα ε, με βία και με ένα ένα όπλο σε ένα έτσι πολύ τρομακτικό βίντεο. Εκατοντάδες κόσμος διαμαρτυρήθηκαν και στο Twitter, αλλά δεν το κατέβασαν και δεν υπήρχε βάση για να το κατεβάσουν από ό,τι φαίνεται. Αν είχε γίνει αυτό στο δρόμο, εγώ θα μπορούσα να το είχα αναφέρει στην αστυνομία, θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι. Αλλά είναι θέμα κλειδί να θυμόμαστε ότι είναι ένας ιδιωτικός χώρος, ιδιωτική εταιρεία που δεν ε, ε, δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Αυτή τη στιγμή το Facebook αρνείται να απαντήσει στην εθνική μας κυβέρνηση. <laughs> αρνείται να έρθει στη Βρετανία να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις για το τι έγινε στο, στο δημοψήφισμα. Είστε οι μόνοι στον κόσμο που έχετε την ε, εξουσία και την αρμοδιότητα και το κύρος να πάρετε απαντήσεις από τον, τον διευθυντή του Facebook και πραγματικά πρέπει να το κάνετε. Και τώρα από την ΑΦΚΟ και το ΕΛΚ η κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, πρώην επίτροπος βεβαίως. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρώην επίτροπος. Ναι, Βεβαίω ε, θα συμφωνήσω και εγώ πως το θέμα του Γενικού Κανονισμού είναι ακριβώς η εφαρμογή που θα έχει και ο ρόλος των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκθεση που θα δημοσιεύσετε στο τέλος του μηνός όπως είπατε αλλά επειδή βλέπουμε ότι η Cambridge Analytica είναι από ό,τι φαίνεται η κορφή του παγωβουνού, αναρωτιέμαι εάν και άλλες αρχές προστασίας δεδομένων ε, σε άλλα κράτη-μέλη κάνουν το ίδιο για να δουν το τι συμβαίνει στην χώρα τους, γιατί πρέπει να λάβουμε δράση στα πολιτικά μας κόμματα για να σωθεί η εκλογική διαδικασία νομίζω πραγματικά κινδυνεύει. Μια έκθεση λοιπόν όπως η δική σας μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν πρέπει να αφορά μόνο την Βρετανία. Πρέπει να γίνει υπό την αιγίδα και των άλλων θεσμικών εποπτών δεδομένων. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η έρευνα αυτή γίνεται λόγω της ε, σχέσης με τη Βρετανία. Και προφανώς οι πόροι μας, γιατί έχουμε πολλούς πόρους, ε, μας ε, επιτρέπουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και εξήγησε και ο συνάδελφός μου το προσωπικό που έχει αφιερωθεί σε αυτή την έρευνα. Λίγες αρχές εποπτείας προσωπικών δεδομένων ε, μπορούν να αφιερώσουν 40 άτομα συν εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες ε, για να ασχοληθούν με τέτοια ζητήματα. Θα σας έλεγα λοιπόν να φροντίσετε οι αρχές προστασία δεδομένων στα κράτη-μέλη σας να είναι επαρκώς στελεχωμένες. Οι συστάσεις της έκθεσής μας θα μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύουν και για παρόμοιες εταιρείε και για παρόμοια κράτη-μέλη. Και βεβαίω ε, θα συνεργαστούμε και με τις πλατφόρμες και με τα κοινωνικά μέσα. Ε, είναι μια καλή χρήση των πόρων μας, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι μια βρετανική μόνο έκθεση, γιατί εστιάζεται στο facebook, στα, στις εταιρείε ανάλυσης δεδομένων, στους μεσίτες δεδομένων, στις ε, προεκλογικές εκστρατείες και τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω λοιπόν ότι έχει ευρύτερη εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Ναι, ναι σημαντικό αυτό. Αυτά συνέβησαν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σαφώς τα μάθη, τα διδάγματα πρέπει να είναι ευρύτερα. Σας ευχαριστώ που το είπατε. Και θα φανεί αυτό και στις επόμενες ακροάσεις. Έχουμε πέντε ομιλητές και η διερμηνία τελειώνει 8. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την βοήθεια των ε, διερμηνέων. Εάν όμως διακοπεί η θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Λοιπόν, ο κύριος Τίμογον από την Γιούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ να απευθυνθώ στον κύριο Παρακύλας. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι το Facebook επιτρέπει στους κατασκευαστές συσκευών πρόσβαση στα δεδομένα. Οπότε από ό,τι φαίνεται γνωρίζουμε μόνο την κορφή του παγόβουνου. Γι' αυτό ανησυχώ. Οι γραπτές απαντήσεις δείχνουν ότι το Facebook θεωρεί ότι η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Facebook και WhatsApp θα είναι αναγκαία στο μέλλον και επιπλέον το Facebook λέει ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές όπως το Flickr, το Vimeo ή το Widget, η διάσημη αυτή η ευρωπαϊκή εφαρμογή. Θεωρείται ότι αυτές οι υπηρεσίες επαρκούν για να οδηγήσουν στην υπόθεση ότι το Facebook δεν έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και θεωρείται ότι αυστηρότεροι κανόνες διαλειτουργικότητας θα βοηθούσαν ή θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η θεωρειτε οτι ειναι παρα πολυ ισχυρη θεση του Facebook και πρέπει να σπάσει το μονοπόλιο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω πρώτα το κομμάτι για τις συσκευές και μετά για το μονοπόλιο σε σχέση με αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα. Η New York Times έβγαλε μια ιστορία σήμερα, ένα ρεπορτάζ και απεκάλυψαν ότι επί σειρά ετών υπήρχε συνεργασία του Facebook με κατασκευαστές συσκευών Samsung, Microsoft, Apple, όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές και στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών προσέφεραν πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς αυτό να είναι σαφές για τους καταναλωτές και επίσης δεδομένα φύλων. Και σε κάποιες περιπτώσεις αποθηκευνούν τα δεδομένα όχι μόνο στις συσκευέ αλλά και στους ε, σερβερ των ε, εταιριών αυτών. Οπότε αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Στις ΕΠΑ υπάρχει το διάταγμα περί συνένεσης της Ομοσπονδιακής ε, Επιτροπής Εμπορίου που απαγορεύει κάτι τέτοιο και δεύτερον Φαίνεται ότι αυτό αντιβαίνει με τα όσα κατέθεσε το ίδιο το Facebook στο Κογκρέσο και αλλού δημοσίως ότι έχει τελειώσει αυτή η άδεια περί δεδομένων φύλων το 2015. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να παρακολουθήσετε στενά την υπόθεση. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι η ιδανική λύση θα ήταν να χωριστεί το προϊόν του Facebook, δηλαδή το Facebook, WhatsApp, Instagram, είτε σε χωριστές εταιρείες, είτε σε εταιρείες που δεν θα μοιράζονται δεδομένα. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή. Παραδείγματο χάρη, αν το γίνεται με το Snapchat, αμερικανική εταιρεία που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το Facebook. Έχουν αντιγράψει τα χαρακτηριστικά του και μετά βεβαίως έπεσε η χρήση του. Ευχαριστώ. Ελκ και Λίβε Τζερόμ Λέναρτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τους κατασκευαστές, αλλά απαντήθηκαν. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κάτι που δεν κατάλαβα και μετά τις ακροάσεις που κάναμε και στο Κογκρέσο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφορά αυτά τα σκιώδη προφίλ, τα shadow profiles. Ο Μαρκ Ζούκερμπερκ μας είπε ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες και για τους μη χρήστες για να λειτουργούν τα προγραμματά μας. Είναι και θέμα ασφαλείας ε, για την ιστοσελίδα μας, αλλά ήταν ασαφής. Δεν μας είπε τι ακριβώς πληροφορίες συλλέγουν. Για μένα δηλαδή, τι είναι, ε, λίστες επαφών, φωτογραφίες, γιατί είναι απαραίτητα αυτά τα στοιχεία για να συνεχίσει να λειτουργεί το Facebook. Ε, αρνήθηκαν ότι δημιουργούν ψεύτικα προφίλ. Αλλά συμφώνησαν, είπαν ότι ναι, παραδέχτηκαν, ε, λαμβάνουν κάποια στοιχεία ε, και ότι εγώ ως μη χρήστη μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και να τα αφαιρέσω. Πώς λειτουργεί αυτό κατά την άποψή σας πρακτικά ε, χωρίς να έχει δημιουργηθεί προφίλ θεωρείτε ότι ισχύει αυτό, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν έχω εγώ επιχειρη... Ε, ε, από πρώτο χέρι ε, από τότε που ήμουν στο facebook για συλλογή δεδομένων από μη χρήστε, αλλά ο κύριος Ζοκερμπεργκ έχει δίκιο. Η συλλογή δεδομένων μη χρηστών είναι πολύτιμη από άψη ασφαλεία για οποιαδήποτε εταιρεία. έχει μια τεράστια ευρεία υπηρεσία διαδικτυακή. Αφορά και τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου. Πολλές στάνταρ τεχνολογίες λειτουργούν έτσι. Δεδομένου αυτών, ε, ο βασικός τομέας ε, όμως που, όπου δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται είναι ότι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ένας χρήστης να επιλέξει να μην συλλεχθούν τα δεδομένα του στο πλαίσιο αυτό ή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά που συλλέξαν, που συνελέξαν και να τα διαγράψει, αν το επιθυμεί. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση το γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι επιλογές διαθέσιμες για τους μη χρήστες. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ε, αυτές οι υποθέσεις γιατί και οι χρήστες και οι μη χρήστες θα πρέπει να έχουν εξίσου τα ίδια δικαιώματα πιστεύω. Ευχαριστούμε για την Λίμπε και Σοσιαλιστέ, η κυρία Άννα Γκόμες. Όπως ανέφερα έχει τελειώσει η δερμηνία να μιλήσετε μόνο αγγλικά.